colleagues, I would Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί κάθεστε εκεί, δεν βρίσκετε θέση. Αν δεν ε, καθίσει κανείς εντός μισής ώρας, μπορείτε να καθίσετε. Καθίστε λοιπόν, αν έρθει κάποιος, μπορείτε να, την, να του δώσετε τη θέση, αν πρόκειται για ευρωβουλευτή, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση για σήμερα, τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Να σα ενημερώσω ότι θα σα πω αργότερα τα, τη συνεδρίαση των συντονιστών αργότερα, προ το τέλος της συνεδρίασης, να ξεκινήσουμε με την έκρηση τη ημερήσια διάταξη. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Νταν Πρέντα ε, ζήτησε την αλλαγή. Μετά από τα σημεία 3 και 4 λοιπόν, θα συζητήσουμε το σημείο 7 και μετά τα σημεία 5 και 6. Το σημείο 7 λοιπόν, το σημείο του κύριου Νταν Πρέντα, θα γίνει μετά από το σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει κάποιο αίτημα αλλαγή, κάποια αντίρρηση. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη και περνάμε απευθεία στο σημείο 2 της ημερήσια διάταξης, που είναι η ακρόαση. Με τίτλο Brexit, συνταγματικέ προκλήσεις και συνέπειες. Ε, για όσους από εσά δεν παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ΑΦΚΟ, ε, να σας πω ότι έγινε ήδη μια συζήτηση, δεν ξέρω αν ήταν στις 16, στις 17, μια ακρόαση. Ε, έχουμε λοιπόν κάνει πάρα πολλή δουλειά την τελευταία χρονιά και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια ε, όσον αφορά τις συνταγματικές πτυχές ε, του Brexit και ως γεγονός και ως διαδικασία. Και για να τα συζητήσουμε όλα αυτά έχουμε προσκαλέσει τρεις εμπειρογνώμονες. Τον καθηγητή Σιώναντα Γκλασκότ, ο οποίος θα μιλήσει για τη ε, διαδικασία της διαπραγμάτευσης ε, για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συνταγματική διάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε τον καθηγητή Πιτ Εκχάουτ για το πεδίο εφαρμογής της ε, Συμφωνίας Αποχώρησης, το θεσμικό πλαίσιο στις συνθήκες, θέματα που αφορούν την ασφάλεια δικαίου, την εφαρμογή και το μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Και έχουμε και τον καθηγητή Κρίστον Χίλιον, ο οποίος θα μιλήσει για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τις σχέσεις μεταξύ της αποχώρησης και της μελλοντική σχέσης και τη συμφωνία που θα έχουμε εκεί, την φύση και την νομική βάση των μεταβατικών μέτρων. Ε, ζητάμε από τον κάθε πυρογνώμονα να αφιερώσει 15 λεπτά στην εισαγωγή του. Προτείνουμε να μιλήσετε με αυτή τη σειρά. Αν θεωρείτε όμως ότι θα μπορούσατε να μιλήσετε με διαφορετική σειρά, δεν υπάρχει πρόβλημα από πλευρά μας. Αν θέλετε να μην μας έχουμε, να δώσουμε πρώτα το λόγο στον καθηγητή Ντάγκλα Σκότ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ την καθηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την πρόσκληση εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στις Βρυξέλλες. Θα, θα μιλήσω αποκλειστικά ε, σχεδόν και μόνο ε, για το συνταγματικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου και το Brexit. Θα σας αναφέρω γενικότερα την ε, κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και το σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και θα πω και λίγα πράγματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, για τη Σκοτία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Καταρχάς, λοιπόν, προφανώς ε, υπάρχει πολύ μεγάλη δουλειά για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για τιτάνιο έργο. Ξέρουμε ότι οι συζητήσεις ε, της αποχώρησης είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή και θα πρέπει καταρχά να καλύψουμε το διαζύγιο, την αποχώρηση αυτή καθ' αυτή και δεύτερον ένα πλαίσιο για μια μελλοντική ε, συμφωνία εμπορίου και ίσως κάποιων άλλων πραγμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον ε, κάποιες μεταβατικές διατάξεις, ε, κάτι το οποίο φαίνεται να γίνεται το ένα και πιο σημαντικό. Ήδη βέβαια ο χρόνος πιέζει και υπάρχει ε, το εξής πάρα πολύ σημαντικό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο να μεταφραστεί σε εγχώριο δίκαιο και να δούμε και τυχόν συνταγματικά ζητήματα και θέματα εκφόρησης ε, εξουσίας και σχέσεις που είχαμε στο παρελθόν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα δηλαδή τα οποία μπορεί να προκύψουν λόγω του Brexit. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι τιτάνιο το έργο πραγματικά και δεν ξέρουμε κατά πόσον θα τα καταφέρουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τούδε. Ε, ο Υπουργό Ορμόδιο για τον Brexit, ο David Davis, ε, πέραν από τι διαπραγματεύσει με τον Μισελ Μπαρνιέ, τι οποίε ξεκίνησε χθε, ε, βγήκε και στο ραδιόφωνο στο Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάνω από 100 σελίδε με λεπτομέρειε ε, για τα σχέδιά του, το οποίο ακούγεται εντυπωσιακό μεν όταν συνειδητοποιήσει ότι αυτέ οι 100 σελίδε είναι απλώς κάποια χαρτιά ε, τα οποία έγραψε το, ε, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Φεβρουάριο για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεύτερον ε, για το πώς θα προκύψει ένα σχέδιο νόμου για την ανάκληση και επίσης για την ομιλία της Τερέζα Μέη στο Lancaster House και φυσικά τα έγγραφα για την αποχώρηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο δηλαδή αυτή τη στιγμή το, η πρώτη λευκή βίβλος ε, πριν από το νομοσχέδιο για την αποχώρηση είναι απλώς κάποιες φιλοδοξίες και η δεύτερη λευκή βίβλος ε, για ε, το σχέδιο νόμου ανάκλησης και πάλι δεν έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Οι νομικοί και άλλοι εμπειρογνώμονες, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω και τον όρο, ε, από τότε που διεξήχθη το δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώνουν ότι και προειδοποιούν ότι υπάρχουν πάρα πολύ πολύπλοκα θέματα σε νομικό και συνταγματικό επίπεδο. Εγώ δεν βλέπω κάπου ότι η κυβέρνηση του Νομένου Βασιλείου είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για αυτά. Θα υπάρχει κόστος για τις δημόσιες υπηρεσίες. Είχαμε και μια περιττή εκλογική αναμέτρηση και προεκλογική εκστρατεία. Και φυσικά ε, Χάσαμε και δύο ε, πολύ σημαντικά μέλη, ε, η Τερέζα Μέη αμέσως μετά τις εκλογές. Το Λόρτ Lord ο, ε, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ήταν αυτός ο οποίος προχωρούσε νομοθεσία για το Brexit στο κοινοβούλιο του Westminster. Και θεώρησε ότι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει άλλο. Και θεωρώ ότι αυτή είναι πάρα πολύ ανησυχητική προοπτική. Στη Σκοτία ε, είμαι ειδική σύμβουλος ε, για τη σκοτική βολή στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων και ξέρουμε ότι η Σκοτία έχει τηρήσει διαφορετική στάση για το Brexit. Η Νίκολα Στέρτζον, ε, Πρωθυπουργό τη Σκωτία στι εκλογέ τη 13η Ιουνίου είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τη θέση της Σκωτία και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ε, συμμετοχή τη Σκωτία και των υπολείπων χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ε, διαπραγμάτευση για τον Brexit. Ε, δεν ξέρω όμω αν ήταν παρόντε και η Πρωθυπουργό τη Σκωτία ή αντίστοιχα οι αρχέ τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Ουαλία στι συζητήσει για τον Brexit. Το θέμα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται θέμα εξωτερικών υποθέσεων, δηλαδή είναι θέμα εσωτερικό, δεν υπάρχει εκχώρηση ε, στις ε, ε, τοπικές βουλές, μπορεί να υπάρχει κάποια διαβούλευση, αλλά δεν μπορούν να έχουν γέννη συμμετοχή. Τώρα, τι γίνεται για, με τις συνέπειες των εκλογών. Η Πρωθυπουργός έχασε την πλειοψηφία της, Ε, από νωρί σήμερα το πρωί βέβαια δεν έχω μπει στο διαδίκτυο, μπορεί να υπήρξαν κάποιες εξελίξεις, αλλά την τελευταία φορά που ε, εξέτασα τα θέματα δεν υπήρξε καμία επιβεβαίωση ότι το DUP θα υποστηρίξει την ε, κυβέρνηση. αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ομιλία τη Βασίλισσας λογικά θα πρέπει να δοθεί στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας και θα ακυρωθεί την επόμενη χρονιά, που αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται ότι είναι πάρα πολύ νομοθεσία που θα πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο τη ε, ε, Westminster και ότι δεν θα πρέπει το 2018 να υπάρξει απέτηση για νέα ε, κοινοβουλευτική ε, συνεδρίαση και να έχουμε ομιλία της Βασίλισσας. Ξέρουμε ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει, πρέπει να υπάρξει μάλλον νομοσχέδιο για να ε, προετοιμάσουμε τη Βρετανία για να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκεί βεβαίω ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία συγγνώμη, να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του άρθρου 50. Πρέπει επίση και όλη αυτή η διαδικασία να περάσει στο εσωτερικό δίκαιο. Αλλιώ θα υπάρξει σωρία προβλημάτων για ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα υπάρχουν κενά, διότι η ε, μεγάλο τμήμα τη Ευρωπαϊκής ε, Νομοθεσίας ισχύει άμεσα, επομένως δεν υπάρχει δική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για το ίδιο θέμα. Ορισμένε φορές πρόκειται για παράγωγο δίκαιο ή δίκαιο το οποίο εκχωρεί εξουσίες και η αρχική πράξη προσχώρηση το 1972 στη, του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις πάψει να ισχύει, σημαίνει ότι πάβει να ισχύει και όλο το παράγωγο δίκαιο. Σημαίνει δηλαδή ότι χάνεται πολύ μεγάλο τμήμα της νομοθεσίας και θα πρέπει να προετοιμαστούμε κάπως γι' αυτό. Αυτό φυσικά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και με ε, κυβέρνηση χωρίς πλειοψηφία δεν θα υπάρχει, ε, θα υπάρχει μάλλον μεγαλύτερο περιθώριο για ε, τροπολογίες της αντιπολίτευσης. Ο Τζέριμι Κόρμπιν, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει πεθάνει το σχετικό νομοσχέδιο. Δεν μπορεί βέβαια να γίνει αυτό, διότι πρέπει να προετοιμαστεί η κυβέρνηση για το πώς θα αποχωρήσει εσωτερικά το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι πρέπει να έχουμε, αλλά σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο περιθώριο για κατάθεση τροπολογιών, για ψηφοφορίες και βεβαίως ε, ε, και η Βουλή των Λόρδων, η Άννη Βουλή, θα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε κρίσιμους τομείς ε, που αφορούν κυρίως δικαιώματα. Δικαιώματα εργαζομένων, κοινωνικά δικαιώματα, ε, για τα οποία έχουμε πολύ, ε, αντλήσει πολλά πράγματα από το ευρωπαϊκό δίκαιο στο εσωτερικό μας δίκαιο και φυσικά έχουμε πει ότι υπάρχει ανησυχία από αυτό. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει εσωτερικώς είναι και ε, το περιθώριο που θα έχουν ε, οι υπουργοί, η εκτελεστική εξουσία, να κάνουν αλλαγές, ε, να ανακαλέσουν νομοθεσία, να τροποποιήσουν νομοθεσία μέσω υπουργικών διαταγμάτων. Ε, ο φόβος ε, που ελοχεύει είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούν ε, να καταργήσουν ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω υπουργικού διατάγματος και αυτό φυσικά σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει μεγάλο περιθώριο συμμετοχής του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Και αυτό θεωρώ είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και το έχουν επισημάνει και αρκετοί για αυτό το νομοσχέδιο. Ε, σε γενικές γραμμές λοιπόν, ε, σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλά ανησυχητικά στοιχεία. Να πω δύο λόγια για να ολοκληρώσω για τη Σκοτία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Και οι δύο χώρες φυσικά ψήφισαν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκοτία με 62% και η σκοτική κυβέρνηση ε, δημοσίευσε και μια λευκή βίβλο με, για τη θέση της Σκωτίας στην Ευρώπη το Δεκέμβριο του 2016, ζητώντας συνεχή ε, συμμετοχή στην ε, νέα αγορά για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ε, εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, τότε απλώς και μόνο για τη σκοτία. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βέβαια ε, δεν ε, έδειξε διατεθειμένη να απαντήσει στη συγκεκριμένη πρόταση γιατί η Πρωθυπουργό δεν το ανέφερε καθόλου στην ομιλία της στο Lancaster House και ε, έκτοτε φαίνεται ότι ξεχάστηκε. Και φυσικά αυτό σημαίνει ότι έμεινε και λίγο περιθώριο για την Σκοτία να προστατεύσει τα συμφέροντά της για την αποχώρηση αλλά θα υπάρξουν σαφώς και συνέπειες ε, για τη συμφωνία ε, ε, για την εκχώρηση εξουσιών, η οποία θα είναι σε μεγάλο βαθμό συνταγματικού χαρακτήρα. Τέλος, αντίθετα, η Βόρεια Ιρλανδία, που είχε 56% υπέρ του Remain, Ε, έχει τύχει αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και από την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείται ότι υπάρχουν ιδιαίτερε μοναδικές συνθήκες και αναφέρθηκε και από την κυβέρνηση, από την Πρωθυπουργό Μέη στην επιστολή ε, για την ε, ε, έναρξη των διαδικασιών του άρθρου 50 και φυσικά είναι και ένα από αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν διαπραγμάτευση αμέσω. Και βεβαίω η ιστορία λόγω των προβλημάτων στη Βόρεια Ιρλανδία και φυσικά στη συνέχεια η ειρηνευτική διαδικασία εν μέρη εξηγούν γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία για τη συγκεκριμένη περιοχή και ιδίω διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να βοηθήσει να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Υπήρξε αναφορά στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και στην κυβέρνηση τη Δημοκρατία τη Ιρλανδία, που είναι και οι δύο μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρονται συχνά στη Συμφωνία τη μεγάλη παρασκευή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδία. Το θέμα είναι τι να κάνουμε. Όλοι λένε ότι δεν θέλουν σκληρά σύνορα μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και της ε, Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Αλλά πώς θα επιληθεί το θέμα αυτό. Δεν είναι ε, αρκετό να έχει απλώς κανείς καλές προθέσεις. Ε, θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση για τη Βόρεια Ιρλανδία από ό,τι φαίνεται, ε, να υπάρχει κάποια μορφή συμμετοχή στην ενιαγορά αγορά και ίσως και κάποια ειδική ρύθμιση για την Τελωνιακή Ένωση, ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα ακριβώ αυτό το σύνορο. Τώρα, το πώ θα το διαχειριστούν όλο αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, διότι αφενός αν θέλεις ε, πιο ε, ανοιχτά σύνορα, δεν θέλεις να υπάρχουν τελειωνιακές ρυθμίσεις, δεν θέλεις να υπάρχουν ε, έλεγχοι διαβατηρίων κλπ. και προσώπων. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να πει να γίνονται έλεγχοι κάπου αλλού. Κάποιο πρότεινε και στην θάλασσα της Ιρλανδίας. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει σύνορο μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και του υπόλοιπου Ηνωμένου Βασιλείου. αλλά η Ατλαντική Ένωση που υποστηρίζει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι δεν θέλει ξεχωριστή μεταχείριση για τη Βόρεια Ιρλανδία σε σχέση με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είμαι λοιπόν βέβαιη πώς θα επιληθεί το συγκεκριμένο ε, ζήτημα. Εάν επιληθεί, τότε και η Σκοτία θα μπορούσε στη συνέχεια να πει ότι ε, θα μπορούσαν να υπάρχουν και ειδικέ ρυθμίσεις για την Βόρεια Ιρλανδία, γιατί όχι και για τη Σκοτία. Και φυσικά η σκοτική κυβέρνηση έχει πολλά στατιστικά στοιχεία τα οποία θα τη βοηθήσουν ε, να επιχειρηματολογήσει υπέρ του γεγονότος ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή απώλεια της ενιαίας αγοράς και θα ήθελαν τουλάχιστον να διατηρήσουν αυτή. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά συνταγματικά προβλήματα για το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit και εδώ και πάρα πολύ καιρό λέω ότι έχω την αίσθηση ότι το Brexit ε, πέραν του γεγονότος ότι ανακλά και τη φύση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει και πάρα πολλά για ε, το συνταγματικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου και ε, τα προβλήματα που έχουμε με αυτές το ευέλικτο μη κωδικοποιημένο σύνταγμα, διότι βλέπουμε ότι ε, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα συνταγματικά εργαλεία για να λύσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, καθηγητά Πιτ Έτκουτ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ευγενή σας πρόσκληση, μεγάλο προνόμιο για μένα να μπορώ να παρίσταμαι εκ νέου στο Κοινοβούλιο για να πω μερικά λόγια για το Brexit. Ετοίμασα και κάποιες διαφάνειες. Δεν είμαι σίγουρος ότι φαίνονται ακόμα στην οθόνη. Εν πάση περιπτώσει μου ζητήθηκε να μιλήσω γενικά για τρία ζητήματα. Το πεδίο εφαρμογή συμφωνία απόσυρση, ποιο είναι ο ρόλο των διαφόρων θεσμικών οργάνων και οι διαπραγματεύσει για την απόσυρση και το θέμα ασφαλείας δικαίου και της υλοποίηση της εφαρμογής μιας ε, ε, συμφωνίας απόσυσης και το μηχανισμό διευθέτησης των διαφορών. Αυτό που θα πω σε μεγάλο βαθμό βασίζεται επί έρευνας που πραγματοποίησαμε συνάδελφο και συντάξαμε και ένα μόλις δημοσιευθέν έγγραφο με αναθεώρηση του, με την Ελένη Φράντζιου για την ε, νομολογία της ενιαίας αγοράς. Είναι ένα έγγραφο για την ερμηνεία του άρθρου 50 από πλευρά συνταγματολόγου. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ανάλυση των διαφόρων διαστάσεων της διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας Απόσυσης δεν καθορίζεται επαρκώ το άρθρο 50, μιλάει για μια συμφωνία για απόσυρση που θα λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων χωρί να λέει τίποτα περισσότερο. Θα γνωρίζετε όλοι, πιστεύω, τις, τους διαπραγματευτικούς προσανατολισμούς που δείχνει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας απόσυρσης. Τα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την απόσυρση είναι θέματα οριζοντίου αρμοδιότητας, που καλύπτουν διαφόρους τομείς νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν θα πρέπει η συμφωνία να επηρεάζει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών μελών. Και γίνεται μια γενική διάκριση μεταξύ της συμφωνίας περί αποσύρσεως και ασδήποτε συμφωνίας για τις μελλοντικές σχέσεις, είτε είναι εμπορική συμφωνία αυτή, είτε μια συμφωνία περί ενιαίας αγοράς ή συμφωνία σύνδεσης. Πιστεύω ότι όσο κανείς αναλύει τις διακρίσεις αυτές, τόσο πιο επισφαλής φαίνεται η όλη προσέγγιση. Μια συμφωνία απόσυρσης πραγματικά αφορά θέματα διαζυγίου του ΣΥΠΗΝ, κληρονομιάς του ΣΥΠΗΝ. Αλλά όλα αυτά καταραίουν σε περαιτέρω ανάλυση. Η συμφωνία απόσυρσης θα τεθεί σε ισχύ τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ πριν από αυτή τη χρονική στιγμή. Κατά κάποια έννοια, διευθετεί και το θέμα των μελλοντικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως όταν γίνεται τη χώρα πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Άκουσα μια άποψη σύμφωνα με την οποία η συμφωνία από ΣΥΡΣΟΣ είναι μια ειδικού τύπου συμφωνία που πρέπει να είναι ξεχωριστή και αρμοδιότητα που δίνει σε αυτή τη συμφωνία το άρθρο 50 πρέπει να είναι διακριτή από την αρμοδιότητα εφαρμογή κοινών εμπορικών πολιτικών και συνάψεω εμπορικών συμφωνιών. η εμπορική συμφωνία μπορεί να συναφθεί με τρίτη χώρα μόνο, αλλά δεν βλέπω μεγάλη διαφορά με τη συμφωνία απόσυρση, διότι και αυτή ε, βασίζεται επί τη ε, προσεγγίσεω σύμφωνα την οποία γίνεται τρίτη χώρα πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να δούμε και ποια είναι η πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Θα καλύπτει αυτή η συμφωνία απόσυρση. Ποια θα είναι τα δικαιώματα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπω υποφαινόμενο, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα, και ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών του Ε.Β. Βασιλείου που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα μπορούσε κανεί όλα αυτά να τα ομαδοποιήσει υπό τον τίτλο Κεκτημένα δικαιώματα. Μπορεί να σκεφτεί και άλλα κεκτημένα δικαιώματα που υπάρχουν. Μια τράπεζα των ΗΠΑ που έχει θηγατρική στο Λονδίνο και εκεί εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά. Αυτή η τράπεζα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι συναισθήθη μια εποχή που ανήκε στην ενιαία αγορά του Ηνωμένο Βασίλειο και έχει κεκτημένα δικαιώματα, Συνεπώ, που θα πρέπει να συνεχίσει να μπορεί να τα απολαμβάνει αυτά τα δικαιώματα. Άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών όσον αφορά το τι θα μπορεί να ρυθμίζει μια συμφωνία απόσυρση. Ξέρω ότι αυτή είναι η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή, διαφοροποίηση μεταξύ διευθετήσεων για απόσυρση και ρυθμίσεως από την άλλη της μελλοντικής σχέσεως. Σαν πολιτική θέση, αν διατηρηθεί αυτή, αν συμφωνήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή θα είναι η προσέγγιση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο να συνδυάσουμε και την απόσυρση και τις μελλοντικέ σχέσεις και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 50 που αναφέρεται απλώς την απόσυρση παραμένουν αρκετά περιθώρια για να ρυθμιστούν οι μελλοντικέ σχέσεις σύμφωνα με το άρθρο 50. Οτιδήποτε συνεχίζει την παρούσα συνεργασία, το παρόν πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ως κάτω μέλος του Ηνωμένου τώρα, αλλά αν παραμείνει στη Europol το Ηνωμένο Βασίλειο, Φερρυπίν, ή αν εξακολουθεί να ανήκει, να καλύπτεται το ευρωπαϊκό ένταμα σύλληψη. Αν συμμετέχει στι πολιτικέ, θα μπορούσε αυτό να ενταχθεί σε μια ενιαία διαπραγμάτευση και μια, σε μια ενιαία συμφωνία. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι η δυνάμη του άρθρου 50 δεν μπορεί καν να διαπραγματευτεί πλήρως τις μελλοντικέ σχέσεις, διότι φαίνεται ότι πρέπει να γίνει κάποια διάκριση σύμφωνα με τα θέματα φορών απόσυρση από τη μια και μελλοντικέ σχέσει από την άλλη, σύμφωνα με το άρθρο 50. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εμπειρία με διεθνεί συμφωνίε με πάνω από μία νομική βάση. Άρα έχουμε μια συνήθιστη ιδέα τώρα που εξετάζουμε, θα μπορούσε να είναι δυνατόν στο τέλος όλα να ενταχθούν σε μία συμφωνία. Σαν νομική βάση, Φερρυπίν, να έχουμε το άρθρο 50 και η εμπορική πολιτική να καλύπτεται από αυτό για τις αρμοδιότητες και αν θέλουμε κάπου σε ευρύτερο πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως τότε θα μπορούσε να έχουμε τη νομική βάση για συμφωνίες συνδέσεως που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαζί με το άρθρο 50 σαν νομική βάση. Βέβαια αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις διαπραγματεύτικέ εντολές για την ώρα που αφορά τα κεκτημένα δικαιώματα, χρηματοπιστωτικά θέματα και θέματα αγοράς, αλλά μπορεί όλα αυτά να εξελιχθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν φύση ως εμπόδια. Όσον αφορά τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων, δεν θα πω πολλά για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου διαπραγματεύσεις. Είναι μια συνηθισμένη ρύθμιση που γνωρίζουμε και από άλλου τομεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε διαπραγματευτική εντολή προς ανατολισμούς από το Συμβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συνάψει τη συμφωνία στο τέλος. Με βάση αυτό, ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου ίσως να ενδιαφέρει και να ανησυχεί. Σημείωσα ότι το Ευρωκοινοβούλιο αυτό κάθε αυτό δεν θεωρείται σαν μέρος των διαπραγματεύσεων σας, διαπραγματεύσει τον Brexit. Είμαι σίγουρος ότι η άποψη του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να εκπροσωπείται στις διαπραγματεύσεις. Θα με ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο τέλος της όλης διαδικασίας, όταν θα υπάρχει μια συμφωνία. Και στο έγγραφο που δημοσιεύσαμε, επιχειρηματολογούμε λέγοντας, και κάτι που θα ίσχυε και το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης, λέμε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι η σύμφωνη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου που απαιτείται για την έγκριση της συμφωνίας απόσυρσης είναι πραγματική σύμφωνη γνώμη αν το προϊόν είναι ένα προϊόν που πρέπει να το δεχτείς να το απορρίψεις και αν η άρνηση συμφώνου γνώμης για τη συμφωνία σημαίνει ότι θα φύγει χωρίς συμφωνία το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε βέβαια μια διετή προθεσμία, αλλά θεωρώ σαν νομικός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 50 και ίσως καμιά φορά να δίνουμε πολύ περιοριστική ερμηνεία στο άρθρο αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι ένας συνταγματολόγος το άρθρο 50 το ερμηνεύει με έναν τρόπο που υποστηρίζει την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα θα πρέπει να προσπαθεί να συνάπτει συμφωνία με το εξερχόμενο κράτος μέλος είναι προτιμότερο παρά να μην υπάρχει συμφωνία. Αυτή είναι συνταγματική απέτηση. Αν το κράτος που αποχωρεί δεν επιθυμεί συμφωνία, δεν υπάρχει λύση. Όμως, αν υπήρξε θέμα διαπραγματεύσεως, μη συμφωνία έχει υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις για κάποια τμήματα συμφωνίας, ακόμα και με μια προθεσμία που επικρέμεται, θα μπορούν διαπραγματευτές να επιστρέψουν στο διαπραγματευτικό τραπέζι και να δώσουν μια νέα συμφωνία η οποία ανατύχει της, συνενέσεως της ε, του Ευρωκοινοβουλίου. Βασίζεται στις ε, δημοκρατικές αρχές η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μοναδική συμφωνία λόγω της διετούς προθεσμίας. Αν αρνηθεί τη σύμφωνη γνώμη το Κοινοβούλιο όπως έκανε για κάποιες διεθνείς συμφωνίες κατά το παρελθόν, δεν συμβαίνει τίποτα, διότι η συμφωνία δεν τίθεται σε ισχύ και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω έκανε ήδη κατά το παρελθόν, ούτω ώστε να ληφθεί υπόψη η ανησυχία του Κοινοβουλίου, μετά επανυποβάλλεται στο Κοινοβούλιο. Σε αυτή την περίπτωση φαίνονται διαφορετικά τα πράγματα λόγω τη διετού προθεσμία. Άρα, εάν γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να αποχωρήσει χωρί συμφωνία το Ηνωμένο Βασίλειο. Και από πλευρά Ηνωμένου Βασιλείου, το συνταγματικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου έχει διευκρινίσει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει και να κυρώσει μια συμφωνία αποχωρήσεως. Να πω τώρα και ποιος είναι ο ρόλος, ενδεχόμενος ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εκεί τίθεται παρόμοια ζητήματα. Δεν βλέπω κάποιο λόγο για τον οποίο δεν θα ήταν εφικτό κάποιο κράτο μέλο ή το θεσμικό αυτό όργανο ή το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, μέλος η γνωμοδότηση του Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού όσον αφορά τη συμβατότητα της συμφωνίας με τις συνθήκες. Η παρούσα νομική θέση είναι ότι το αίτημα για γνωμοδότηση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και το δικαστήριο ποτέ δεν δέχτηκε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά θα υπάρξει μια υποχρέωση που θα επιβάλλεται στα άλλα θεσμικά όργανα και στον Ηνωμένο Βασίλειο να περιμένουν για, το, για την απόφαση του δικαστηρίου πριν ε, εφαρμόσουν και ολοκληρώσουν τη διεργασία, τη συμφωνία. Να πω ένα-δύο πράγματα για την ασφάλεια δικαίου, επιβολή, διευθέτηση διαφορών στα πλαίσια συμφωνίας απόσυρσης, δηλαδή να δημιουργηθεί κλίμα ασφαλείας δικαίου, όταν τίθεται σε ισχύ η συμφωνία απόσυρση εξορισμού του Ηνωμένου Βασίλειου τρίτη χώρα και δεν θα ισχύουν πλέον για τη χώρα αυτή ε, συνθήκε. Αλλιώ δεν είναι συμφωνία βάσει του άρθρου 50 για να δημιουργήσει, για να έχει συνέπεια αυτή η συμφωνία για την νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να ενταχθεί στην νομοθεσία, να ενσωματωθεί στην νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάποτε διαβάζω κάποιε ανησυχίε που εκφράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το σεβασμό του, των όρων της συμφωνία αποσύρσεω. Πρέπει να πω ότι αν αυτά ενσωματωθούν στην Εθνική Νομοθεσία, τα δικαστήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο σίγουρα θα στηρίξουν την εφαρμογή των όρων μια τέτοια συμφωνία, για να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου και κυρίως σκέφτομαι το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών και από τις δύο πλευρές, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν χρήσιμο αυτή η συμφωνία να έχει άμεση ισχύ όσον αφορά την νόμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή να μπορεί να επιβληθεί ε, σε οποιοδήποτε δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στη συμφωνία. Αυτή καθ' αυτή η διαπραγματική εντολή και οι οδηγίες αναφέρονται σε ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποσύσεως. Εκεί όλος ιδιαίτερος αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτή είναι μια πρόταση άνευ Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα παραδείγματα περιπτώσεων όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει γενική δικαιοδοσία όσον αφορά θέματα που αφορούν νομοθεσία ενός ε, μη κράτου μέλους, όπως θα θεωρείται μετά την απόσυση του Ηνωμένου Βασίλειου, και με πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι άνθρωποι όπως εγώ, που διαμένουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, έχουμε καλυμμένα τα δικαιώματά μα και μπορούμε να αποσφύγουμε στο ΔΕΚ. Ο μόνος δρόμο να φτάσουμε εκεί θα είναι η προδικαστική απόφαση, ούτω ώστε να μπορούν τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου να υποβάλουν ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό προϋποθέτει όμως συμμετοχή με άμεση εφαρμογή του, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ότι είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις του ΔΕΚ στα εσωτερικά δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου επικράτηση του ευρωπαϊκού δικαίου και δεν μπορώ να δω πώς θα γίνει αυτό να εφαρμοστεί στην νομοθεσία μιας τρίτης χώρας που δεν θα καλύπτεται πλέον από ε, τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχω κάποιες αμφιβολίες για το πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει στην πρακτική και κατά πόσο μάλιστα θα συμφωνεί το Ηνωμένο Βασίλειο με κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρχει, ρόλο, υπάρχει κάποιος ρόλος για το ΔΕΚ, μπορεί να εφαρμοστεί συμφωνία απόσυρσης. Πώς ρυθμίζονται οι διαφορές μπορούμε να έχουμε ένα μοντέλο διαθέτηση των διαφορών που είναι διακυβερνητική μορφής. Πολύ πιο δύσκολο να έχουμε ένα μοντέλο που θα εμπλέκει και ιδιωτικά, ιδιωτικούς φορείς, πολίτες, οι εταιρείε, ή νομικά πρόσωπα να μπορούν να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δικαστήριο τύπου ΕΖΕΣ. Ξέρω ότι αυτό ε, προτάθηκε, ότι θα μπορεί να γίνει μέλος της ΕΖΕΣ τελικά και να γίνει μέλος του δικαστηρίου της ΕΖΕΣ στο Ηνωμένο Βασίλειο, άρα θα υπάρχει ένας θεσμός που θα μπορούσε να λειτουργήσει. Να το πάρουμε αυτό σαν πρότυπο, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Το δικαστήριο ΕΖΕΣ έχει πάνω από ένα δικαστή ε, και δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που διευκρίνησε ότι δεν ήταν δυνατό να έχουμε ένα δικαστήριο ΕΟΧ με δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από την πλευρά και, από, και δικαστές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου την άλλη. Το μοντέλο ΕΖΕΣ, του δικαστηρίου του ΕΖΕΣ, είναι ένα εξωτερικό μοντέλο. Και προδικαστικές αποφάσεις, αν είναι δυνατόν το δικαστήριο ΕΖΕΣ να προχωρήσει σε αυτό το πεδίο, πώς θα λειτουργούσε, να δημιουργηθεί ένα ειδικό δικαστήριο για τους σκοπούς αποφάσεως επί διαφορών όσον αφορά την συμφωνία απόσυρση, δεν ξέρω αν θα λειτουργούσε και έχουμε ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο σήμερα όσον αφορά η αντίποτε συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε μορφές διευθετήσεως διεθνών διαφορών. Είναι το θέμα της αυτονομίας του, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής που τονίζει το ΔΕΚ όλος ιδιαίτερος στην πρόσφατη νομολογία του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βασικά στα πορίσματα περί πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βασίζεται επί της αρχής του δικαστηρίου, σύμφωνα την οποία κανένας φορέας διευθετήσεως, διεθνής, διεθνής φορέας διευθυντής διαφορών θα μπορούσε να ερμηνεύσει την ομολογία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν έχουμε συμφωνία απόσυρσης που όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών της Εμπλοκής Ενώσεως στο Ενωμένο Βασίλειο θέλει να διατηρήσει τα ισχύοντα δικαιώματα σύμφωνα με την Ομοθεσία της Εμπλοκής Ενώσεως, αυτό προβλέπουν οι διαπραγματικές οδηγίες, να διαφυλαχτούν αυτά τα δικαιώματα στο βαθμό του δυνατού, τότε αναπόφευκτα οτιδήποτε δικαστήριο θα πρέπει να δει πώς θα ερμηνεύσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ούτως ώστε να εφαρμόσει μια τέτοια συμφωνία. Τώρα, αν αυτό θα δεχτεί την ευλογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν ξέρω, διότι έχει μια ευρεία ερμηνεία της αυτονομίας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και με τις εμπορικές σχέσεις δημιουργούνται δύσκολα προβλήματα όσον αφορά τη διευθέτηση των διαφορών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Κριστό Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας για την πρόσκληση μου ζητήθηκε να εξετάσω διάφορες πλευρές της ε, διαπραγματευτικής διαδικασίας από συνταγματική πλευρά. Λόγω του περισμένου χρόνου θα περιοριστώ σε τρία θέματα. Το πρώτο είναι μια επενθύμηση. Η διαδικασία αυτή δεν καλύπτεται μόνο από τη διαδικασία του άρθρου 50, αλλά περιορίζεται επίσης και γενικότερα από τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Δεύτερον, η εφαρμογή του άρθρου 50 ήδη είχε ως αποτέλεσμα την ε, εκπόνηση και περαιτέρω κανόνων και αρχών πέρα από το στενό περιεχόμενο του άρθρου 50 που επίσης θα παίξουν ρόλο στη διαδικασία αποχώρησης. Και το ένα θέμα είναι οι φάσεις της ε, διαδικασίας και το ενδεχόμενο εφαρμογής μεταβατικών διακανονισμών. όλα αυτά τα αναφέρουν οι επιπλέον κανόνες. Ε, αυτοί οι κανόνες είναι ένα αναδιόμενο ε, αποχωρησιακό δίκαιο και ορισμένες φορές δεν συνάδουν με το άρθρο 50. Και το τρίτο που θα αναλύσω αν έχω χρόνο είναι να επισημάνω τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ρόλο του στη διαδικασία αποχώρησης. Λοιπόν, υπενθυμίζω τη σημασία του Ευρωπαϊκού Σταματικού Δικαίου για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Όπως ξέρετε, το άρθρο 50 αναφέρει δύο βασικές προϋποθέσεις για την διαπραγμάτευση. Πρώτον, ποιος είναι ο στόχος. Συγκεκριμένα, να συμφωνηθούν οι ρυθμίσεις για την αποχώρηση και να διαμορφωθεί πλαίσιο για τις περαιτέρω μελλοντικέ σχέσεις του αποχωρούντος κράτους με, το, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερον, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, να συμφωνήσει για μια συμφωνία μετά την έξοδο, μετά τον Brexit. Και αυτή είναι η θέση που νομίζω ότι υιοθέτησε και χθε σε ένα βαθμό και η Βρετανική αντιπροσωπεία, από ό,τι κατάλαβα. Το δεύτερο στοιχείο του άρθρου 50 είναι το διαδικαστικό πλαίσιο για την διαπραγμάτευση της συμφωνίας αποχώρησης. Καθιστά σαφές στο άρθρο 50 ότι οι διαπραγματεύσεις είναι στα χέρια των ενωσιακών θεσμών. Αντίθετα με την ενταξιακή διαδικασία που είναι στα χέρια των κρατών μελών, τουλάχιστον τυπικά, η διαδικασία αποχώρησης είναι αρμοδιότητα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από την Ένωση και όχι τα κράτη-μέλη. Η συμμετοχή των ενωσιακών θεσμών σε μια διαδικασία κοινοτικού τύπου. Θα δείτε ότι χρειάζεται, για παράδειγμα, ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο για την ολοκλήρωση τη συμφωνία, χρειάζεται συμφωνή γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το δικαστήριο μπορεί να παίξει ρόλο. Αυτή η κοινοτική μέθοδος και η συμμετοχή των θεσμών σημαίνει ότι η διαδικασία αποχώρησης είναι ε, σαφώς εντός του ευρωπαϊκού συνταγματικού πλαισίου είναι ενταγμένη εκεί. Αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσει δεν θα πρέπει να γίνουν μόνο με βάση το άρθρο 50, αλλά και τηρώντα του βασικού κανόνε συνταγματικού ενωσιακού δικαίου. Και αυτό έχει διάφορε επιπτώσει. Να αναφέρω μερικέ. Πρώτον, οι διαπραγματεύσει πρέπει να γίνουν με πλήρη τήρηση του γενικότερου πλαίσιου λειτουργίας τον θεσμό της Ένωσης. Για παράδειγμα, το άρθρο 13, όπως έχει ερμηνευθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεύτερον, οι θεσμοί πρέπει να δρουν με, σε συμφωνία με τους κανόνες για την ε, κατανομή αρμοδιοτήτων και εντός της Ένωσης και εντός των ενωσιακών θεσμών αλλά και μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών. Άρα υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των ε, διαπραγματεύσεων αποχώρησης και των διαπραγματεύσεων για την κατάσταση μετά την Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμφωνήσει, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί μία συμφωνία για σχέσεις με ένα κράτος μέλος όταν αποχωρεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις εμπορικές του σχέσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση. Επίσης, Η διαδικασία αυτή γίνεται με βάση και τις βασικές λειτουργίες των θεσμών. Δηλαδή, να βοηθάει την Ένωση να επιτυγχάνει τους στόχους και να εκτελεί τα καθήκοντά της. Όπως αναφέρει το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προωθεί τις αξίες της, να, εξετάζει, να φροντίζει για την ευημερία των ε, πολιτών της και γενικότερα περαιτέρω προβλέψεις του άρθρου αυτού. Δηλαδή, οι θεσμοί, ενώ διαπραγματεύονται τη διαδικασία αποχώρηση όσο και αν φαίνεται παράδοξο, θα πρέπει να βοηθούν την Ένωση να προωθεί την ενοποίησή της. Διαπραγματευόμενοι λοιπόν την συμφωνία αποχώρησης, οι θεσμοί, όχι πρέπει μόνο να σεβαστούν τις ε, θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, την αρχή της μη διάκρισης για παράδειγμα, θα πρέπει να διατηρήσουν και την ακεραιότητα της νομικής τάξης και τις τέσσερις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει να διατηρούν και το κεκτημένο στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Όλες αυτές οι αρχές κάπως ε, αντανακλώνται στις κατευθύνες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και, ε, στην ε, οδηγία και στις διαπραγματεύσεις. Καθορίζουν τι μπορεί να κάνει η Ένωση στα πλαίσια της διαδικασίας αποχώρησης και τι δεν μπορεί να κάνει. Άρα καθορίζουν και τον βαθμό ευελιξίας που έχει η Ένωση στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης. Καθορίζουν τι μπορεί να συμφωνήσει η Ένωση με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά με τις διαπραγματεύσεις μιας ε, κλασικής ε, εξωτερικής ε, συμφωνίας όπου υπάρχει πολύ περισσότερο περιθώριο για δούνε και λαβίν. Γιατί το κράτος μέλος στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας παραμένει μέλος μέχρι να αποχωρήσει. Και σε αυτά το πλαίσιο και αυτό το λέει επανειλημμένα το κείμενο των ε, κατευθυντηρίων γραμμών, το Ευρωπαϊκό, συγγνώμη, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις ε, υποχρεώσεις του ως μέλος της Ένωσης, για παράδειγμα, από την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας. Άρα δεν μπορούν να δράσουν μεμονωμένα τα κράτη-μέλη στους τομείς που καλύπτει η διαπραγματευτική διαδικασία. Οι καθημερινές γραμμές είναι σαφείς σε αυτό και ιδιαίτερα κατηγορηματικές. Δεν μπορούν να κάνουν ad hoc συζητήσεις για θέματα που αφορούν την διαπραγματευτική διαδικασία. Άρα τα χέρια της Ένωσης και των κρατών μελών είναι δεμένα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει καθόλου περιθώριο για ευέλικτες, ε, ευέλικτους διακανονισμούς. Για παράδειγμα, διατηρώντας την ε, ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς, η Ένωση μπορεί να πρέπει να προτείνει νέους διακανονισμούς γιατί η ενιαία αγορά δεν περιορίζεται σε 27 κράτη-μέλη, περιλαμβάνει και τρεις χώρες ΕΖΕΣ. Ό,τι συμφωνηθεί μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου για τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο παράλληλα να εφαρμοστεί και για τον χώρο ΕΖΕΣ. Πρέπει λοιπόν κάπως να συμμετάσχουν και οι χώρες ΕΖΕΣ. Αν όχι στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία διατήρησης της ακαιρεότητας της εσωτερικής αγοράς και σχεδιάζοντας μεταβατικές ε, ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεύτερο σημείο τώρα, που ακριβώς ε, σχετίζεται με τη δυνατότητα ευέλικτων ρυθμίσεων στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης παρά το ότι είναι δεμένα τα χέρια της Ένωσης. Το άρθρο 50 και τώρα το ανακαλύπτουμε. Δεν καλύπτει όλες τις πλευρές της ε, διαδικασίας αποχώρησης. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Γι' αυτό χρειάζονται επιπλέον κανόνες και αρχές. Αυτό μας φέρνει στην σταδιακή ανάπτυξη των ε, κανόνων διεύρυνση της Ένωσης που βασίζονταν και στο άρθρο 49 αλλά και πέρα από αυτό για να οργανωθεί η ένταξη νέων μελών. Μέχρι στιγμή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βασίζεται στο άρθρο 50 όπως δείχνουν και οι κατευθυντήρες γραμμές του. Δύο παραδείγματα να αναφέρω. Μεταβατικές ρυθμίσεις και η αλληλουχία των φάσεων της διαπραγμάτευσης. Η αλληλουχία δεν λέγεται πουθενά εκπεφρασμένα στο άρθρο 50. Με ποια σειρά θα πρέπει να γίνουν οι διαπραγματεύσεις αποχώρησης. Ίσως υπάρχει έμεσα μία αναφορά στο ότι πρώτα πρέπει να γίνει αποχώρηση και μετά η μελλοντική σχέση. Αλλά δεν αναφέρεται σαφώς. Η πρώτη φάση θα εστιάσει στο να δώσει ασφάλεια για τους κύριους εμπλεκομένους και να διασφαλίσει την αποδόμηση των σχέσεων των δύο πλευρών. Μας λένε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει πότε θα θεωρήσει ότι έχει επιτευχθεί επαρκή πρόοδο σε αυτή την πρώτη φάση, ούτω ώστε οι διαπραγματεύσει αποχώρηση να περάσουν στη δεύτερη φάση, όπου οι δύο πλευρέ θα έχουν προπαρασκευαστικέ και προκαταρκτικέ συζητήσει για τι μελλοντικέ του σχέσει. Όπω και στην διαδικασία ένταξη παρατηρούμε μία ε, αλληλεξάρτηση των δύο φάσεων της διαπραγμάτευσης. Και αυτό θέτει θέμα για την συμβατότητα αυτής της αλληλεξάρτησης με τους όρους και το στόχο του άρθρου 50. Ιδιαίτερα, οι κατευθυντήρες γραμμές δεν εξηγούν ιδιαίτερα τι σημαίνει υπαρκής πρόοδος. Δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια. Πότε οι διαπραγματεύσεις μπορούν να περάσουν στη δεύτερη φάση. Αυτό επαφείται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κατά πάσα πιθανότητα με ομοφωνία. Με συνένεση. Αν και έχει επίσης ε, αναφερθεί ότι ο κύριος Μπαρνιέ θα μπορούσε να παίξει βασικό ρόλο. Λοιπόν, αν θεωρηθεί ότι υπάρχει επαρκής πρόοδος, συγγνώμη, αν δεν υπάρξει επαρκή πρόοδο, μπορεί να κολλήσουν οι πραγματεύσει. Δηλαδή, ένα κράτο μέλο, ένα μόνο κράτο μέλο θα μπορούσε να πει εγώ δεν θεωρώ ότι έχει υπάρξει επαρκής πρόοδο. Δηλαδή, επανέρχεται το βέτο. Φεύγουμε λοιπόν από την κοινοτική μέθοδο, που ήταν μια πολύ ενοποιημένη, μια πολύ ενιαία διαδικασία. Βεβαίω είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η κοινοτική μέθοδος για να καθοριστούν οι προτεραιότητες που τι ανέφερε και ο Πιτ. Αλλά αυτή η σταδιακή προσέγγιση, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εκλεπτυνθεί περαιτέρω για να δούμε τι κριτήρια θα, θα έχουμε ως βάση και για να αποφευθεί αυτή η δυνατότητα ένα κράτος μέλος για εσωτερικού λόγου, για παράδειγμα, όπω έχει γίνει τόσες φορές πρόσφατα, στα πλαίσια της διαδικασίας διεύρυνση, ένα κράτος μέλος λοιπόν να μπορεί να εκβιάζει και να μπλοκάρει τη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σεβαστέ οι ευρύτερε συνταγματικέ αρχές. Και ίσως έτσι κάπως να αλλάξουμε και τη θεσμική ισορροπία που αρχικά προέβλεπε το άρθρο 50. Τώρα, μεταβατικές ρυθμίσει. μας είπαν ότι θα συμφωνηθούν στα πλαίσια της δεύτερης φάσης με βάση ένα νέο σύνολο διαπραγματευτικών οδηγιών που θα προτείνει υποθέτω η Κομισιόν και θα κρίνει το Συμβούλιο. Λέγεται ακόμη ότι θα γίνει κάτι τέτοιο μόνο εφόσον είναι προς το συμφέρον της Ένωσης και για να δημιουργήσουμε γέφυρες για τη μελλοντική σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε, υπάρχουν καλοί, σκόπιμοι λόγοι για να υπάρξουν μεταβατικέ ε, ρυθμίσει. Αλλά όπω και με τη σταδιακή προσέγγιση, με την προσέγγιση δηλαδή από τη μία φάση σε δύο φάσει, μπορεί να θέσουν νομικά θέματα, ιδιαίτερα σε σχέση με το άρθρο 50. Ένα θέμα συγκεκριμένο. Και είναι ένα μόνο από τα θέματα. Δεν είναι σαφέ αν αυτέ οι μεταβατικέ ρυθμίσει και μέτρα θα πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν σε ένα χωριστό πλαίσιο ή αν θα συμπεριληφθούν στην συμφωνία αποχώρησης. Η ταπεινή μου γνώμη. Θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην συμφωνία αποχώρησης. Στο κείμενό της. Εάν βέβαια, διότι υποθούν έτσι, ούτως ώστε να είναι αναγκαίες για τους σκοπούς της αποχώρησης. Δηλαδή, εάν στηρίζουν την όλη διαδικασία αποχώρησης θα μπορούσαν να συμπεριφθούν στη συμφωνία. Γιατί θα ε, ήταν επιβοηθητικές του κυρίου στόχου που είναι να καθοριστούν οι όροι της αποχώρησης. Ο Πιτ είπε ποια ήταν η ερμηνεία της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την ε, κοινοτική αρμοδιότητα που βασίζεται στο άρθρο 50 και που είναι οριζόντια και καλύπτει τα πάντα. Ο τρόπος που καθορίζεται και ερμηνεύεται αυτή η διάταξη επίσης θα στήριζε αυτή την άποψη ότι η Συμφωνία Αποχώρησης θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα μεταβατικά μέτρα όσο ευρεία κλίμακα και αν είναι. Αλλά μπορούμε να επανέλθουμε στη συζήτηση. Γιατί πολλά βέβαια εξαρτώνται από το περιεχόμενο. Και το στόχο αυτών των μεταβατικών μέτρων. Υπάρχει όμως κάτι σαφές. Αυτές οι μεταβατικές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να έχουν ως στόχο να προκαθορίζουν τη μελλοντική σχέση των δύο πλευρών. Υπάρχει ένα θεματολόγιο σύνδεσης στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας για να εφαρμοστεί ακόμη επικείμενη συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία. Η έννοια της ε, φάσης εφαρμογής κατεμένα σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι διαπραγματεύσει για τη μελλοντική σχέση να συμφωνηθούν στα πλαίσια αυτής της διετούς περίοδου και ότι στην ουσία θα ήταν ε, η όρη εφαρμογή μια νέα εταιρική σχέση κατόπιν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια του άρθρου 50 κατά τη γνώμη μου. Τέλο, τέλο. Δύο λεπτά να αναφέρω τι σημαίνουν όλα αυτά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το άρθρο 50 υπενθυμίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να δώσει σύμφωνη γνώμη για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και επειδή η διαδικασία μπορεί ε, το επιτρέπει, μπορεί το Κοινοβούλιο να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να ζητήσει μια γνώμη για τη συμβατότητα με το νοσιακό δίκαιο της συμφωνίας, αλλά για να αμφισβητήσει κάποιο νομικά δεσμευτικό μέτρο στα πλαίσια της διαδικασίας. Επειδή θα μπορούσε να αναδείξει στις συνθήκε αυτό το μέτρο. Για να μπορέσει να ασκήσει δικαστικό έλεγχο το Κοινοβούλιο. Άρα έχει πολλές δυνατότητες το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και μπορεί και να αξιοποιήσει και την ομολογία του δικαστηρίου για θέματα θεσμική ισορροπία στα πλαίσια του άρθρου 218, το οποίο και αυτό συμμετέχει στη διαπραγματεύση. Για παράδειγμα, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να έχει πλήρη πληροφόρηση με βάση για τα τεκτενόμενα, με βάση την ομολογία. Οπότε θα σας πρότεινα δύο συγκεκριμένα που μπορείτε να κάνετε ως κοινοβούλιο. Πρώτον, να επαγρενείτε πάντα για να ελέγχετε ότι τηρούνται οι βασικές συνταγματικές αρχές από τους συμβαλωμένους στη διαπραγμάτευση. Την Επιτροπή δηλαδή και το Συμβούλιο μέσω της Ομάδας Εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επαγρυπνεί και να ελέγχει. Ούτως ώστε να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό αυτών των συνταγματικών αρχών από τους διαπραγματευόμενους. Εάν υπάρχει λοιπόν μια διαπραγμάτευση με δύο φάσεις, σε δύο φάσεις, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε να μην μπορεί να μπλοκάρει το Συμβούλιο ή κάποιο κράτος μέλος στη διαδικασία. Ένα δεύτερο καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Α, έλειξε ο χρόνος μου. το Κοινοβούλιο θα μπορούσε ακριβώς να βοηθήσει στην εκπόνηση των κριτηρίων για το τι σημαίνει επαρκής πρόοδος για να πυροδοτηθεί η δεύτερη φάση. Έχει μέσα, με βάση το άρθρο 50, έχει όπλα, αλλά και γενικότερα. Έχει και ένα γενικότερο λόγο. Το Κοινοβούλιο είναι το μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο από πλευρά Ένωση που συμμετέχει στη διαδικασία. Άρα αυτό νομιμοποιεί την πρόθεσή του να παίξει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σέπφλιν. Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει με τους συντονιστές, θα δούμε τους υπόλοιπους. Ο Τζόρτζ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τις, τους τρεις ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Προς την καθηγήτρια Ντάγκλα Σκότ ε, απευθύνει τη ερώτησή μου. Η φύση του συντάγματος του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν ξέρω αν ακούτε, η φύση του συντάγματος του Ηνωμένου Βασιλείου Τα μελέτησα αυτά πριν από πάρα πολύ καιρό και γνωρίζω κάποιες συμβάσεις του συντάγματος, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο απουσιάζει είναι οποιαδήποτε συνδεδεμένη νομοθεσία. Το σύστημα το οποίο πορεύει από τη σύμβαση του Ντάισις είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει αποτέλεσμα όταν μπορεί να εφαρμοστεί αυτοπεριορισμός. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρχει μια σοβαρή διαταραχή στο σύστημα, λειτουργεί ομαλά. Και νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια διπλή διαταραχή. Μία είναι το μέλλον της Σκοτίας. Ποιο θα είναι το μέλλον της Σκοτίας ε, σε αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο ε, είτε ανεξάρτητο είτε μη ανεξάρτητο και πάλι θα υπάρχει πρόβλημα διότι ουσιαστικά αποτελεί ξεχωριστή μονάδα. Και ε, ε, τι σχέση θα έχει με το Λονδίνο και βεβαίως ε, δευτεροβόντως το Brexit. Θεωρώ ότι αν τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, σε κάποιο βαθμό έρεται ο παραδοσιακός αυτοπεριορισμός και δεν ξέρω αν είμαι πάρα πολύ αυστηρός εδώ, από πλευράς κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ουσιαστικά υπάρχει δυνατότητα να δρά ευθέρετα τροποντινά, αυθαίρετα την Να λαμβάνει αποφάσεις, ε, δεν υπάρχει κατεπίγουσα νομοθεσία, αλλά η κυβέρνηση συμπεριφέρεται ε, σαν να βρισκόμαστε σε μια κατεπίγουσα κατάσταση. Και η ερώτησή μου είναι εάν μπορεί να υπάρξει κάποια ρύθμιση στη συνταγματική τάξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως σε κάποια χρονική στιγμή μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Brexit. Γιατί αν όχι, τι εταίρος θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η Mercedes Πρέσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, στην επίλυση διαφορών. Αν ε, κατάλαβα καλά, διότι αντιμετωπίζουμε πάντα μια πάρα πολύ περίπλοκη κατάσταση, ε, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ελβετίας, που θα μπορούσε να είναι και ένα πιθανό ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το δικαστήριο αποφαίνεται μεν, αλλά Στη συνέχεια υπάρχει θεσμικό όργανο στην Ελβετία, δεν ξέρω ακριβώς ποιο, το οποίο ε, αποδέχεται ουσιαστικά την απόφαση. Πρόκειται λοιπόν για μια μορφή συμφωνία, ε, μέσω της οποίας αποφασίζει με το δικαστήριο, αλλά από εκεί και πέρα γίνεται ε, μια διαδικασία ε, παραλαβής ουσιαστικά της απόφασης. Ε, δεν είναι αυτόματη αυτή η διαδικασία. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα. Όλες οι υπόλοιπε μου φαίνονται αδύνατες σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εκτός και αν υπάρξει κάποια διεθνή συνθήκη και χρησιμοποιηθεί αυτή, αλλά τότε θα πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Το δεύτερο ζήτημα αφορά το γεγονός ότι αρκετοί από εσάς αναφέρθηκαν στα στάδια της διαπραγμάτευσης. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε διάφορα στάδια διαπραγμάτευσης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η συμφωνία δεν θα προβλέπει, όπως προβλέπει και το άρθρο 50, τη συμφωνία αποχώρησης και το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων. Και επομένως και από πλευράς ε, ψήφου, η ψήφο θα είναι πάλι η ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 50, γιατί εν τέλει η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα πράγματα. Επομένως δεν ε, βλέπω με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετική ε, δυνατότητα ψηφοφορίας, να υπάρχει και ομοφενία και ειδική πλειοψηφία. Νομίζω ότι αυτό διευκρινίζεται από το άρθρο 50. Και μια πολύ σύντομη ερώτηση για το πώς ερμηνεύετε εσείς τη μεταβατική συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι είναι απλώς αυτό που συμβαίνει μεταξύ της επίσημης αποχώρησης και της μελλοντική συμφωνίας. Δηλαδή αυτό το διάστημα που έχει τελείως διαφορετικό ε, καθεστώς, ισχύει διαφορετικό δίκαιο και φυσικά τα χρονικά είναι τελείως διαφορετικά. Ε, για μένα λοιπόν αυτή η μεταβατική συμφωνία θα πρέπει να είναι απλώς ε, το πώς θα συμπεριφέρει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε κάποιο βαθμό, γιατί φυσικά πλήρως ίσως να είναι και δύσκολο, μέχρι την τελική νέα συμφωνία. Το πλαίσιο των σχέσεων βεβαίως είναι ένα πλαίσιο ε, από πραγματική συμμετοχή, για παράδειγμα στην ενιαία αγορά ή σε μια σειρά από άλλα ευρωπαϊκά νομοθετήματα, διότι αν είναι μια συμφωνία η οποία είναι σαν συμφωνία με κράτος μέλος δεν χρειάζονται μεταβατικές διατάξεις. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και από εσά ε, λίγο πώς τη βλέπετε αυτή την πτυχή. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει μόνο εάν στη συμφωνία προβλέπεται και ένα ε, πλαίσιο σχέσεων που δίνει ένα διαφορετικό καθεστώς ε, στη Μεγάλη ε, Βρετανία και δεν θεωρείται απλώς ένα τρίτο ε, κράτος. Υπάρχει δηλαδή συμμετοχή σε μία σειρά από ευρωπαϊκά ε, κεκτημένα, για παράδειγμα την Εννέα αγορά και την τελωνιακή ένωση. Βλέπω μόνο εγώ, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, αλλά θα μπορούσε να είναι και θέματα ασφαλείας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο. Για όλα αυτά σε αυτή την περίπτωση, ε, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει κατά την άποψή σας αυτή η μεταβατική συμφωνία. Ε, συνάδελφοι, έχουμε 11 άτομα που θέλουν να λάβουν το λόγο. Αν θέλετε να ακούσετε και τις απαντήσεις, ε, τρία λεπτά ο καθένας σας παρακαλώ. Ο κύριος Βοιαστός και από το ECR. Παρακαλώ τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω την εντύπωση ότι όλοι υποθέτεται ότι το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Εξού και η ερώτησή μου, ποιες είναι οι προβλέψεις σας, σε ποιες σφαίρες, σε ποιους τομείς το Βρετανικό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει ρόλο ελεγκτικό σε ποιο βαθμό θα αλλάξουν οι απόψει του, Ευρωπαϊκού, του Βρετανικού Κοινοβουλίου με λαμβάνοντα από τι εκλογέ. Τελευταίο από του συντονιστέ, η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Κυρία Σπινέλη, για την ΚΟΥ έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις έξοχες εξηγήσεις σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας και την απεσιοδοξία του καθηγητού του κ. Ντάγκλα Σκότ. Δεν υπάρχει πραγματική προετοιμασία, αυτό πιστεύω, ούτε από πλευράς ενώσεως, ούτε από πλευράς Βρετανικής κυβερνήσεως. Και έχουμε και τα προβλήματα Σκοτίας και Βορείου Ιρλανδίας. Σοβαρά προβλήματα. Έχουμε πολύ λιγότερο από δύο χρόνια στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι ο χρόνος πραγματικά είναι πολύ πιο σύντομος και οι πιθανότητες μη συμφωνίας ε, να αυξάνονται. Εξαρτάται μόνο από την επισφαλή θέση της Βρετανικής κυβερνήσεως ή από την έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επίσης. Γι' αυτό συμφωνώ με την ιδέα του τελευταίου που μίλησε, του καθηγητή Έκχουτ, μάλλον. Αν είναι σύντομο το χρονικό διάστημα και αν υπάρχει κίνδυνος μη συμφωνίας, είναι σημαντικό η μεταβατική συμφωνία να συμπεριληφθεί στη συμφωνία αποχώρησης. Έτσι τουλάχιστον δεν δημιουργείται ένα πλήρες κενό όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και το θέμα της Βορείου Ιρλανδίας. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου. Δηλαδή, να προχωρήσουμε βάσει της αρχής ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι ότου να υπάρχει συμφωνία επί των πάντων. Είναι μια διατύπωση που πάντα μου δημιουργούσε αμφιβολίες. Τι σημαίνει αυτό. Ότι επίσημη και οριστική συμφωνία για τα δικαιώματα των πολιτών ή όσον αφορά την προστασία της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και όσον αφορά το δικαίωμα της Ιρλανδίας να έχει αυτές τις δύο ε, φύσεις αν θέλετε δεν μπορεί να ρυθμιστεί αν δεν λυθούν τα άλλα ζητήματα, μια συμφωνία για τα χρηματοπιστωτικά κλπ. πριν υπάρξει τελική συμφωνία. Μια άλλη ερώτηση. Αναφερθήκατε στην πιθανότητα μιας ε, συμφωνίας τύπου ΕΖΕΣ. Έχω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Προβλέπει η ΕΖΕΣ τις τέσσερις ελευθερίες και την ελευθερία μετακίνησης των προσώπων. Δεν νομίζω ότι αυτό θέλει η Βρετανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον επιθυμία της παρούσης κυβερνήσεως. Θεωρείται ότι θα ήταν δυνατόν. Έστω και σαν υπόθεση εργασίας. Η, η δυνατότητα διαχωρισμού των τεσσάρων ελευθεριών. Έχουμε τρεις ελευθερίες που δίδονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και να μην υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Αυτό το ενδεχόμενο το αναφέρω διότι πρόσφατα κάποιες προσωπικότητες όπως ο καθηγητής Πισανιφέρη ε, σύμβουλος του Μακρόν και κάποιος άλλος ε, Βρετανός βουλευτής του οποίου το όνομα λησμόνησα, πρώην υπουργό ήταν, του Μπλερ, ξέχασα ποιο είναι από το όνομά του, το ανέφεραν αυτό. Άλλη μια ερώτηση, ευχαριστώ Μπάρμπαρα, και μετά θα ζητήσουμε από τους εμπειρογνώμονε να απαντήσουν. Ο κ. Μέσο Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις έξοχες παρουσιάσεις. Θα τηρήσω το τρίλεπτο μου, αλλά έχω μια ερώτηση για κάθε μέλο του πάνελ. Πρώτα, στον κύριο Ντόγκλα Σκοτ. Είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα χάσει τη δευτερογενή νομοθεσία. Δεν το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την πρωτογενή, αλλά τη δευτερογενή με βάση την αμοιβαιότητα όλα θα μπορούσαν με μία πράξη να εφαρμοστούν. Η δυσκολία είναι όταν υπάρχει αμοιβαιότητα μεταξύ των δύο φορέων. Οπότε υπάρχει απέτηση αμοιβαία αναγνώριση. Πολλέ οδηγίε όμω, κανονισμοί και όλα αυτά αποτελούν κανονική νομοθεσία Από την παρόλο των ετών έχουν επικρατήσει τη εθνική νομοθεσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούσε με μια νομοθετική πράξη αυτά να τα διατηρήσει. Οι δυσκολίε που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί να μην εμπνευστεί από τη Γρυλανδία, η οποία ανήκει στο Μεγάλο Βασίλειο τη Δανία, όπω και εγώ, αλλά δεν ανήκει στην αγορά-αγορά. Έφυγε το 1996. Δεν είναι κάποιο παραλληλισμό που θα μπορούσε να γίνει. Γεωγραφικά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Νομικά δεν είναι κάτι παρόμοιο. Κύριε Εκχάουτ, για το θέμα που συζητούσατε για την ΕΖΕΣ. Κάποτε είχα μια υπόθεση μεταξύ κάτω μέλους Ισλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, κάποια διαφορά που υπήρχε. Δεν υπάρχει ανάγκη και τα δύο μέρη σε μια υπόθεση ΕΖΕΣ να είναι μέλη της ΕΖΕΣ αυτής καθεαυτής. Και γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ένα νέο νομικό σύστημα που θα καλύπτει μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφετούνται διαφορέ. Ε, κύριε Σλιόν, είπα, αναφέρατε κάποιε σκέψει για το άρθρο 13 και τις αξίες του άρθρου 3 και συμπεράνατε ότι έτσι καθίσταται ανέφικτη δυνατότητα παραλλήλων διαπραγματεύσεων. Δεν το καταλαβαίνω. Αν το 3.6, άρθρο 3 σημείο 6, που λέει ότι η Ένωση θα επιδιώκει του στόχου τη που προαναφέρονται, με τα δεδειγμένα μέτρα, λαμβάνοντα υπόψη και τι αρμοδιότητε που ανατίθονται από τι συνθήκε. Η ίδια διατύπωση ακριβώ που είχαμε όταν η Γρυλανδία διαπραγματεύτηκε την έξοδό τη και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα τότε. Οι ελευτικέ συμφωνίε με τη Γρυλανδία να, να συνάπτονται όταν είχε εξέλθει και για το ρόλο του Κοινοβουλίου δεν αναφέρεται στο άρθρο 50 του Κοινοβούλιο ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει κάποιο ρόλο, κανένα ρόλο στι διαπραγματεύσει. Λέει ότι θα πρέπει να αποφασίσει και μόνο και αναφορά στο 218, άρθρο 218 σημείο 3, αλλά δεν προβλέπεται εκεί κάποιο ρόλο για το Κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνω από πού προέρχονται όλε αυτέ οι ανησυχίε σα. Ευχαριστώ. Να δώσουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων. Λοιπόν, τέσκαν πολλές και δύσκολες ερωτήσεις. Λοιπόν, με τη σειρά υποβολής και πολλές αφορούσαν τη δική μου ομιλία. Πρώτον, η φύση του συντάγματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ε, εντάξουμε νομοθεσία. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον ε, κατά τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ότι μας επέτρεψε μέσω της ε, συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στη, μέσω του νόμου που εγκρίθηκε για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές κοινότητες να εγκρίνουμε μέτρα. Τώρα θα φύγουμε και θα χάσουμε αυτή τη δυνατότητα να εγγράφουμε μέτρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και όπως σας είπα υπάρχουν δύο απόψεις για το Σύνταγμα. Μία είναι η ιδέα του Ντάισι για την κυριαρχία του Κοινοβουλίου και η άλλη λαμβάνει υπόψη πιο πρόσφατες εξελίξεις της ε, συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη, για το νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της περιφέρειας. Και η ανησυχία είναι ότι θα χαθεί αυτή η δυνατότητα ε, ορισμένοι νόμοι να στηρίζονται σε ευρύτερους ενουσιακούς νόμους. Γιατί αν κρατήσουμε αυτά τα δικαιώματα και γίνουν ε, εθνικοί νόμοι, η παραδοσιακή άποψη για το Σύνταγμά μας ε, δίνει τη δυνατότητα να τα καταργήσει. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την Τζίνα Μίλλερ είπε ότι δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε η εκτελεστική εξουσία. Πρέπει να γίνει μέσω νόμου για να ε, γίνει η επίκληση του άρθρου 50 τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τι θα προκύψει. Ανησυχούσα πάρα πολύ μέχρι ίσως τις, πρόσβατες, τις πρόσφατες εκλογές γιατί από τη μία είδαμε ε, την εθνικιστική άποψη που έλεγε ότι, που έλεγε ότι αυτό που θέλουμε είναι μια ανεξάρτητη Σκοτία και μια ενιαία Ιρλανδία και από την άλλη μεριά ορισμένοι έλεγαν όχι μας αρέσει πώς λειτουργεί το Σύνταγμα και πιστεύουμε στην πρωτοκαθεδρία του Κοινοβουλίου. Κανείς δεν μίλησε για φεντεραλισμό ή για περαιτέρω χώριση αρμοδιών στις περιφέρειες. Δεν ξέρω λοιπόν αν η τελική ρύθμιση θα σημαίνει περαιτέρω Θα το δούμε. Ορισμένα άλλα. Να επανέλθω σε αυτό που είπατε στο τέλος, αλλά γιατί λυπάμαι. Ε, δεν ξέρω αν ε, δεν εκφράστηκα καλά. Τι εννοούσα ως δευτερογενή νομοθεσία. Ήταν η δευτερογενής νομοθεσία στο Ενωμένο, στο Ενωμένο Βασίλειο. Πολύ σημαντική ενωσιακή νόμοι, για παράδειγμα οι κανόνες για το χρόνο εργασίας, έχουν γίνει ε, δευτερογενές δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου και παράγωγο δίκαιο. Και ε, αναφερθήκατε στην κατάσταση το προηγούμενο της ε, ε, Γρυλανδίας. Αυτό υπόθηκε για την περίπτωση της Σκοτίας ε, να γίνει μια αντίστροφη δηλαδή διαδικασία Γρυλανδίας. Δηλαδή ένα τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου η Σκοτία να μείνει και άλλοι να φύγουν. Η παραδοσιακή απάντηση ήταν όχι. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Ε, άλλες οι σχέσεις Γρυλανδίας και Δανίας γιατί στην περίπτωση της αποχώρησης της Γρυλανδίας το κέντρο της χώρας και η πρωτεύουσα έμειναν στην Ένωση. Τι έννοια θα έχει να μείνει η Σκωτία αν φύγει το Λονδίνο και η Αγγλία. Και υπάρχουν πολύ σημαντικές αρμοδιότητες οι οποίες ε, εδράζουν στην, ε, στο Λονδίνο, εξωτερική πολιτική, οικονομική πολιτική, πάρα πολλά. Στην περίπτωση της Γρυλανδίας ήταν πολύ μεγαλύτερη η αυτονομία της Γρυλανδίας. Θα χρειαζόμασταν ένα νέο συνταγματικό διακανονισμό, μια νέα συνταγματική συμφωνία δεν αποκλείεται. Αλλά μέχρι στιγμής αποφεύγει τέτοια συζήτηση η Βρετανική κυβέρνηση. Η ε, περισσότερων, αρμοδιοτήτων, για παράδειγμα, στη Σκοτία και την Ηνωμένα Ιρλανδία και την ε, Βόρεια Ιρλανδία. Αν θέλουμε να λύσουμε, για παράδειγμα, το Ιρλανδικό, θα πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητε στη Βόρεια Ιρλανδία για να μπορέσει να αποφασίσει. Θα πρέπει να γίνουν λοιπόν αλλαγέ. Έγιναν πολλές άλλε ερωτήσει. Ε, ξέρω ότι ο χρόνος περιορισμένος, οπότε θα περιοριστώ. Α, κάτι ακόμη. Τίθενται κάποιε ερωτήσει για το εάν μπορεί το Κοινοβούλιο της Βρετανίας να ψηφίσει επί τη συμφωνία αποχώρησης. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο Πρωθυπουργό είπε ότι θα πρέπει να ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Αλλά τι είναι θα έχει αυτή η ψηφοφορία αν είναι ναι ή όχι. Αν είναι Δηλαδή το δίλημα εάν δεν υπερψηφίσετε αυτή τη συμφωνία θα φύγουμε χωρίς καμία συμφωνία. Ή αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις και πρέπει και πάλι να αποχωρήσει χωρίς συμφωνία. Τι μπορεί να κάνει το Βρετανικό Κοινοβούλιο για να το αποφύγει, για να το αποτρέψει. Μετά τις εκλογές τώρα μοιάζει να υπάρχει πλειοψηφία κατά της άποψης ότι καλύτερα να φύγουμε χωρίς συμφωνία παρά να καταλήξουμε σε μια κακή συμφωνία. Αλλά τώρα τι ακριβώς θα μπορέσει να κάνει το Βρετανικό Κοινοβούλιο για να επιβάλλει την άποψή του δεν μου είναι ακόμη σαφές. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου να κάνω και μια πρόταση σε σχέση με την τελευταία σας παρατήρηση. Βεβαίω και θα ήταν δυνατόν να υπάρξει διαπραγμάτευση μια συμφωνία αποχώρηση, η οποία κυρίως... Ε, θα αφορά και την ε, συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να γίνει αποδεκτή και από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα μπορούσε να το προβλέπει δηλαδή η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ, αυτή τη στιγμή θα έχει εγκριθεί και από τα Κοινοβούλια. Και νομίζω ότι το άρθρο 50 ε, μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα άρθρο το οποίο επιτρέπει και ε, τέτοιους όρους ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τώρα σε σχέση με τις συμφωνίες με την Ελβετία. Εδώ και αρκετό καιρό πιστεύω ότι κάνουμε μια συζήτηση τελείως άσπρο-μαύρο στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, λες και ε, μόνο ένας είναι ο τρόπος για να ε, διαδραματίζει το ρόλο του το δικαστήριο και αν είναι θέματα της δικαιοδοσίας του ή όχι. Η δικαιοδοσία του βεβαίω είναι μία από τις κόκκινες γραμμές μετά από τις πρόσφατες εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα κόκκινη αυτή η γραμμή, άλλαξε λίγο χρώμα αλλά σίγουρα μπορούν να δοθούν νέε απαντήσει ε, στο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για παράδειγμα, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο Ηνωμένο Βασίλειο και το αυτό ισχύει και για το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ε, του ΕΟΧ. Επομένως, είναι τελείως διαφορετική θεσμική θέση σε σχέση με ε, το κατά πόσον ε, προτεύει και το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και βέβαια μπορεί να έχει και ένα πιο ίσονο σημασίας ρόλο και να λέμε ότι βάση της νομολογίας θα λαμβάνεται υπόψη ίσως στη νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, το κατά πόσον μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές συμφωνίες αυτό, θα συμφωνούσε εδώ και εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες από μία συμφωνία, διότι ρυθμίζουμε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη μελλοντική σχέση, παρά το γεγονός ότι δεχόμαστε ότι το άρθρο 50 όλα αυτά τα υποδηλώνει. Και όσον αφορά τη μετάβαση, εγώ δεν είπα τίποτα στην αρχική μου παρέμβαση για τη μεταβατική διαδικασία αλλά ε, κατά την άποψή μου ε, είναι πολύ μεγάλο ε, θέμα και μας ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί σε δύο χρόνια δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε πλήρη διαπραγμάτευση της νέας σχέσης και το πώς θα είναι αυτή η μεταβατική συμφωνία ε, αν δεν έχεις αποφασίσει προς τα που οδεύεις, πώς θα μπορέσεις να έχεις μια πλήρη μετάβαση μέσα αυτής της οδού. Πώς μπορείς να ξέρεις τι εμπορικές σχέσεις θα έχεις στο μέλλον και αν θα υπάρχει πλήρης τελωνιακή ένωση ή τι τελωνιακή ένωση θα υπάρχει ή η συμμετοχή στην ενία αγορά κλπ. Πώς μπορεί να γίνει η συμμετοχη στην ενια αγορα κλπ πως μπορει να γινει η μεταβαση σε κάτι το οποίο είναι ακόμα αβέβαιο ε, για το μέλλον. Εγώ δύο τρόπους βλέπω να γίνει μετάβαση. Από τη μια να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο λίγο περισσότερο και να παραταθεί η διάρκεια του άρθρου 50 ή να έχουμε ένα μοντέλο σαν τον ΕΟΧ, αλλά και αυτό θα είναι δύσκολο διότι αν δεν είναι ο ΕΟΧ αυτός καθεαυτός, αλλά είναι μια συμφωνία που θα είναι αντίστοιχη με τον ΕΟΧ, ε, τότε δεν έχουμε στην πραγματικότητα μια μετάβαση, έχουμε μια πλήρη διαπραγμάτευση για μια πλήρη νέα σχέση. Νομίζω λοιπόν ότι η όλη έννοια της μεταβατικής συμφωνίας ε, είναι αρκετά ε, επισφαλής εδώ. Βεβαίω, ε, θα πρέπει στην συμφωνία απόχώρηση να υπάρξει και διαπραγμάτευση για τη μεταβατική διαδικασία. Όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία και το τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να έχουν συμφωνηθεί τα πάντα, νομίζω ότι το θέμα δεν τίθεται μόνο για τη Βόρεια Ιρλανδία, τίθεται γενικότερα ε, για τα ε, δικαιώματα και ε, ο συνάδελφός μου στο Πανεπιστήμιο όταν αναφέρθηκα και στα Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο και το πρόβλημα που υπάρχει γιατί απασχολούν και πολύ προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν του είπα ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα θεώρησε ότι αυτή είναι η πιο ε, τρομακτική πτυχή της όλης διαπραγμάτευσης. Το να υπάρξει λοιπόν συμφωνία για τα δικαιώματα των πολιτών που θα εφαρμοστούν πριν συμφωνηθεί οτιδήποτε άλλο, κατά την άποψή μου είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις τέσσερις ελευθερίες, να έχουμε μόνο τρεις και όχι τέσσερις από πλευράς νόμου για συμφωνία με τρίτη χώρα που παρέχει μόνο τρεις ε, ελευθερίες και όχι την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εγώ δεν πιστεύω, δεν ξέρω αν έχει άλλη άποψη ο Κριστόφ, ε, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι στο συνταγματικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να το απαγορεύει. Είναι μάλλον μια πολιτική έννοια, ως πολιτική έννοια την αντιλαμβάνουμε πλήρως, διότι εάν ε, προσφέρονται τρεις ελευθερίες και όχι τέσσερις, ε, ε, γιατί να μην ακολουθήσουν και άλλα ε, κράτη-μέλη και να προσπαθήσουν να αποχωρήσουν και αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για συμφωνία με χώρα που δεν είναι μέλος, ίσως θα μπορούσε. Τώρα, για τον κώδικα ΕΖΕΣ και μια τέτοια συμφωνία. Η ανησυχία μου είναι ότι η πρόσβαση ε, από τους πολίτες, ε, ένα δικαστήριο εζές, το αν θα έχουν πρόσβαση πολίτες σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ε, δεν είναι δυνατόν για το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχέση που έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαν μόνο μία πλευρά της όλης διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα λειτουργούσε ένα τέτοιο δικαστήριο ΕΖΕΣ με μόνο μία χώρα, εκτός και αν γίνει δεκτό ότι θα υπάρχουν και Ευρωπαίοι δικαστές ε, σε αυτό το δικαστήριο, που δεν θα είναι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άλλοι δικαστές που θα ε, διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δεχτεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ένα τέτοιο μοντέλο, οψόμεθα, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Καλώς. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Την τελευταία ερώτηση. Άρθρο 13 και άρθρο 36. Τι ήθελα να πω. Στα πλαίσια του άρθρου 50, τα θεσμικά όργανα κινούνται στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Νόμου και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις του άρθρου 13. Το άρθρο 13 έχει δύο πτυχε. Καθορίζει τι εντολέ των θεσμικών οργάνων. Για να πετύχει στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθούνται οι αξίε αυτή κλπ. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 13 προβλέπει ότι οι βασικέ αρχέ που διέπουν τη διάδραση μεταξύ των θεσμικών οργάνων καθορίζουν τα όρια στα οποία κινούνται σέβεται ο μεν τις εξουσίες του άλλου και θα εφαρμόζουν ειλικρινή συνεργασία. Τι προσπαθούσα εγώ να πω. Το θεσμικό στοιχείο θέλω να τονίσω. Όταν θεσμικό όργανο διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμικά όργανα, πρέπει να δρουν εντός των ορίων των εξουσιών τους, τηρώντας πλήρως το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τίποτα στο άρθρο 50 καθορίζει παρέκκληση από αυτή την αρχή. Τα θεσμικά όργανα πρέπει να κινούνται εντός των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί. Άρα πρέπει να σέβονται το Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο περί επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στον τομέα του εμπορίου είναι σαφή τα όρια των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Το εμπόριο είναι εμπορική αποκλειστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τα κράτη-μέλη στο τομέα του εμπορίου μπορεί να κινηθούν αν του δοθεί η έγκριση και άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν του δοθεί τέτοια άδεια, βεβαίω τα κράτη-μέλη θα δρουν σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν μπορεί να του δοθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να του δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξουσία που δεν έχουν για να παραβούν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι λέω με όλα αυτά όσο το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει κράτο μέλο. Και αυτό υπογραμμίζεται πολλέ φορέ στου ανατολισμού και στι οδηγίε για τι διαπραγματεύσει. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να παραβεί το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ενώση, πρέπει να το σέβεται. Καλώ. Άρα, τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα που το Ηνωμένο Βασίλειο σαν κράτο μέλο δεν έχει αρμοδιότητα. Τα θεσμικά όργανα δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα παρέβαιναν τον νόμο. Αυτό ήθελα να πω. Δεν αναφερόμουν στο άρθρο 3.6. Στο άρθρο 3 αναφερό, αναφέρεται στα καθήκοντα που έχει η Ένωση. Η διαπραγματευτική διαδικασία στα πλαίσια του άρθρου 15 οδεύουν επικαθορισμού λεπτομεριών για αποχώρηση κάτω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μια εντολή για επανεξέταση του ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσης εκτός το απολύτως αναγκαίου για τους σκοπούς αποχώρησης. Εγώ ανέφερα το άρθρο 3, διότι ήθελα να πω ότι τα θεσμικά όργανα στις διαπραγματεύσεις δεσμεύονται. Πρέπει να προστατεύσουν το κεκτημένο. Το κεκτημένο μπορεί να τροποποιηθεί στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο για τους σκοπούς διευθετήσεως της αποχωρήσεως. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι αρκετά αυστηρή ερμηνεία, ένα αυστηρά Αυτό ήθελα να πω. Αν επιτρέπετε, για τη Γρυλανδία να πω κάτι. Ήταν εντελώ διαφορετική η κατάσταση η Γρυλανδία. Η Γρυλανδία ποτέ δεν ήταν κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάλογο εκτό μικροφώνου. Δεν ακούνε οι διερμηνεί. Απάντηση. Σαν τμήμα τη Δανία, η Γρυλανδία δεν ήταν ένα ξεχωριστό κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα. Η σύγκριση αυτή, με κάθε σεβασμό για του Βρετανού φίλου μα, η σύγκριση τις περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την περίπτωση της Γρυλανδίας δεν είναι κάτι απόλυτα σωστό, νομικά τουλάχιστον. Η ιδέα ότι η Γρυλανδία μπορούσε να διαπραγματευτεί αλληλευτική ρύθμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ηρώταν από το πεδίο εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στα πλαίσια του συνταγματικού πλαισίου της Δανίας δεν είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για του σκοπούς της συζητήσεως. Θα, θα πρέπει να συζητήσετε περαιτέρω κάτι αυτό γιατί έχουμε και άλλες ε, ερωτήσεις. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι για τις ε, μεταβατικές ρυθμίσεις. Στον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις, λοιπόν, υπόθηκαν αρκετά. Τι πιστεύω εγώ. Οι μεταβατικές ρυθμίσεις, όπως ερμηνεύω εγώ τα πράγματα, υποτίθεται ότι αρχίζει να ισχύει αρχίζουν να ισχύουν τη στιγμή που θα αποχωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έννοια γέφυρα που γεφυρώνει την κατάσταση μέλου Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τη μελλοντική διευθέτηση φαίνεται να είναι ο σκοπός της μεταβατικής ρύθμισης. Αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση στη δεύτερη φάση. Και αυτό τι δείχνει. Ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τουλάχιστον πρότεινε ότι πρέπει αυτό να ανήκει σαν κομμάτι στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων αποχώρησης. Άρα θεωρείται ότι η μεταβατική ρύθμιση θα συμπεριλαμβάνεται στη Συμφωνία Αποχώρησης. Και νομίζω ότι είναι λογικό. Όχι μόνο λόγω του χρονισμού, αλλά και λόγω των όρων που επιβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει του άρθρου 50 και μέσω των διαπραγματευτικών εντολών που ανατέθησαν. Αν θέλουμε μεταβατική ρύθμιση σε ξεχωριστό μέσο, το θέμα τη νομική βάση και του εργαλείου θα τεθούν του μέσου αυτού. Και ποια θα είναι η φύση αυτού. Πρέπει να είναι μεικτό ή όχι. Προβλέπω ότι κάποια μεταβατική διευθέτηση ίσω άπτεται τομέων τη κοινών αρμοδιοτήτων Ευρωπαϊκή Ενώσεως και κρατών μελών. Άρα δεν έχει λόγο να έχουμε ξεχωριστό μέσο, διότι θα είναι εγκαίρω έτοιμο να λειτουργήσει από τη στιγμή που θα έχει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά το περιεχόμενο και το σκοπό, φαντάζομαι ότι ίσω να είναι πολλαπλά αυτά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε σταδιακή εξάλληψη μέτρων. Να γίνει λιγότερη, λιγότερο βία η αποχώρηση σε κάποιου τομεί πρέπει να εντοπιστούν. Το θέμα τη ηθαγένεια ίσω είναι ένα τομέα. ίσως να ακολουθηθεί άλλη προσέγγιση, μη μεταβατική και άλλη τομή ίσως, όπου σταδιακή αποχώρηση θα είναι απαραίτητη. Τώρα, αν θα υπάρχει σταδιακή εφαρμογή και προσέγγιση όσον αφορά τις μελλοντικές ρυθμίσεις, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ μακριά αυτή η προσέγγιση. Καταλαβαίνω αυτό που λες Πιτ ότι δεν μπορεί να έχει κανείς σωστή μεταβατική διευθέτηση όταν δεν γνωρίζει ποια θα είναι η μελλοντική συμφωνία. Εγώ θα έδινα μια άλλη απόχρωση. Αν τα μέρη συμφωνούν ότι θα υπάρξει συμφωνία σύνδεσης με σφαιρική προσέγγιση για το ελεύθερο εμπόριο, έχουμε κάποια ιδέα του αντικείμενου της πραγμάτευσης και θα πρέπει να συζητηθούν στο μέλλον οι λεπτομέρειες. Αν πρόκειται αυτή να είναι η συμφωνία στη δεύτερη φάση μεταξύ των δύο μερών, των διαπραγματεύσεων της συμφωνίας αποχώρησης ότι η μελλοντική σχέση θα είναι μια συμφωνία σύνδεσης ή χώρος ελεύθερου εμπορίου, ο σκοπός της μεταβατικής ρυθμίσεως φαίνεται λογικός. Να μην ξαναδημιουργηθούν εμπορικό εμπόδια τα οποία θα πρέπει να αρθούν εκ νέου όταν θα συναυθεί η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και θα τεθεί σε ισχύ. Εκεί μπορεί να υπάρχει σταδιακή εφαρμογή μέτρων και προσεγγίσεων η μεταβατική ρύθμιση δεν μπορεί να ερμηνευτεί δεν μπορεί να ερμηνευτεί σαν, φάση ε, εφαρμογής μελλοντική συμφωνίας. Πρέπει να ξέρουμε πρώτα ποια θα είναι η μελλοντική κατάσταση πριν ακολουθηθεί αυτή η φάση της εφαρμογής. Τέλος, για τη μεταβατική διευθέτηση. Η συμμετοχή, το θέσατε αυτό για τη συμμετοχή. Εγώ θα το πω ομά. Δεν υπάρχει συμμετοχή κράτους μέλους που δεν είναι πλέον κράτος μέλος. Από τη στιγμή που ένας κράτος μέλος αποχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάνει τα, Συγγνώμη, χάνει τα συμμετοχικά δικαιώματα. Επειδή υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις, δεν υπάρχουν συμμετοχικά δικαιώματα. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Αν το δει αυτό κανείς από τη σκοπιά της ε, Νορβηγίας ε, του Λίχτενστάιν, πώς είναι δυνατόν ένα πρώην κράτος μέλος να έχει κάποια συμμετοχικά δικαιώματα σε μεταβατική διευθέτηση, όταν εμείς που είμαστε μέλος της ε, ε, εσωτερικής αγοράς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο για την εσωτερική αγορά και την ακαιρεότητα των ρυθμίσεων. Και τέλος, οι λέτε τέσσερις ελευθερίες. Δεν γνωρίζω αρκετά από αυτού, αλλά θέτω το θέμα ως εξή. Η ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και εργαζομένων πώς θα λειτουργήσει σαν σήμερα χωρίς ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Δεν το κατανοώ. Θα ήταν άλλου είδους ελευθερίες. Ναι, πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαπραγματευτεί κάποιε κάποιες συμφωνίες με τρίτα κράτη-μέλη για ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και εργαζομένων προχωρούν σε αρκετό βάθος, αλλά δεν μπορεί νομίζω να πάρει μόνο τρεις από τις ελευθερίες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλα αυτά που συνεπάγεται να τα εντάξει σε μια συμφωνία και να αφήσει παράμερα μια ελευθερία. Άρα θα είναι πολύ δυσλειτουργική η όλη έννοια των τεσσάρων ελευθεριών. Είχα αρκετά σημεία και άλλα σημεία που θέλω να θέσω, αλλά έλειξε ο χρόνο μου. Ε, Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Δύο λεπτά παρακαλώ, επόμενοι μιλητέ, γιατί έξι θέλουν να πάρουν το λόγο. Σα παρακαλώ να περιοριστείτε. Richard Corbett. Ευχαριστώ χωριστή συμφωνία για τα δικαιώματα των πολιτών για να αποφύγουμε το πρόβλημα του τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα το συζητήσαμε και έθεσα το ερώτημα στον κύριο Μπαρνιέ που είπε ότι δεν γίνεται απόλυτα έχετε αντίθετη άποψη δεύτερον η άποψη που είπατε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ενιαία συμφωνία με διτή νομική βάση αλλά αν ε, υπάρχει τέτοια συμφωνία, τότε η επικύρωση της συμφωνίας θα αφορούσε και τις δύο πλευρές. Δηλαδή του Εθνικού Κοινοβουλίου για την πλευρά άρθρου 50 αυτής της διαδικασίας. Και αυτό βέβαια θα ήταν πολύ προβληματικό. Τρίτον, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αν το Κοινοβούλιο ή ακόμη και ένα κράτος μέλος προσφύγει κατά της συμφωνίας λέγοντας ότι δεν είναι συμβατή με τις συνθήκες ή με τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είπατε ότι δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μα θα έπρεπε το δικαστήριο, θα έπρεπε να σταματήσει να μετράει ο χρόνος μέχρι να αποφασίσει. Και άρα, λόγω όλων αυτών, δεν υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε ένα ε, εντελώς ε, περιορισμένο ε, διαζύγιο που θα επιλύσει μόνο τα εντελώς στοιχειώδη και οι μεταβατικές ρυθμίσεις θα είναι ότι παραμένει το status quo για 3-4 χρόνια μέχρι να λυθούν όλα τα υπόλοιπα που θα καθορίσουν τη μελλοντική σχέση. Και αυτό δεν θα έθετε σοβαρά θέματα από πλευρά δημοκρατία γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Βρετανικό Κοινοβούλιο θα επεκύρουν συμφωνήσουν που δεν έχουν λύσει κανένα από τα βασικά θέματα που έχουν όλα αναβληθεί. Ο κύριος Φλάναγκαν έχει φύγει. Δεν τον βλέπω. Η Μαρτίν Άντερσον. Σας ευχαριστώ για τις παρουσίες, παρουσιάσεις. Αν θα μπορούσατε να μας στείλετε παρακαλώ. Και οι τρεις. Στην ε, καθηγήτρια Douglas Scott. Με ενδιαφέρουν αυτά που είπατε γιατί το Brexit υπονομεύει τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Και επειδή η συντηρητική κυβέρνηση τελικά δεν κατάφερε το στόχο της μέσω των εκλογών, η θέση του DUP είναι να εδρεώσει τη διχοτόμηση της Ιρλανδίας. Ακούσαμε ένα βουλευτή τους να μας λέει ότι χρειάζονται απολύτως αυστηρά σύνορα. επειδή η συμφωνία της ε, Μεγάλης Πασκευής είναι η διεθνή συμφωνία που έχει κατατεθεί και στα Ηνωμένα Έθνη και δύο κράτη είναι οι συνεγγύητες. Η Βρετανική κυβέρνηση ενώ θα έπρεπε να δράμε απόλυτη αμεροληψία σε σχέση με το Βορρά, όχι πως το κάνει ποτέ, τώρα αποδεικνύει τώρα που κάνει γλύκες με το DUP ότι σίγουρα δεν θα είναι απόλυτα αμερόληπτη για την εφαρμογή της συμφωνίας. Θέλω λοιπόν να καταλάβω το 3.5 που λέει ότι η Ένωση δεν θα διευκολύνει παραβιάσεις διεθνούς δικαίου. Και επειδή η Συμφωνία της Μεγάλης ε, Παρασκευής είναι λοιπόν διεθνή συμφωνία, γι' αυτό βασίζουμε στο 3.5 και στο 8 που λέει ότι η Ένωση μπορεί να έχει μια ειδική σχέση με μια γειτονική περιοχή. Άρα, η πρότασή μας που λέμε ότι θα πρέπει να είναι ειδικό καθεστώς καθορισμένο η Βόρεια Ιρλανδία είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική λύση σε αυτήν ε, την πανολεθρία του Brexit για τις επιπτώσεις που θα έχει για τους πολίτες της Ιρλανδίας και ιδιαίτερα για τους πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας και για το πώς θα θίξει τελικά και τις συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι ευρωβουλευτή ε, του Λονδίνου. Θέλω να μιλήσω ω ευρωβουλευτή του Λονδίνου για το 1 εκατομμύριο του οποίου εκπροσωπώ και το πανεπιστημιακό από το από την εκλογική μου περιφέρεια και υπάρχουν και πάρα πολλοί ενωσιακοί πανεπιστημιακοί. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι Εάν τα προγράμματα των κομμάτων δεσμεύουν την κατάσταση ή αν θα μπορούσε η κυβέρνηση να συνεχίσει την ε, κατάσταση όπου θα συνεχιστεί η σύγκληση μέχρι τη στιγμή της αποχωρήσης και μετά βεβαίως θα υπάρξει απόκληση. η ερωτήσεις μου είναι εξής. Μία είναι με τα κεκτημένα δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης να ψηφίζουν στις τοπικές περιφερειακές εκλογές. Είναι τόσο σημαντικό αυτό για να ακούγεται η φωνή τους, έστω περιορισμένα. Επειδή εκπροσωπώ το Λονδίνο για 18 χρόνια, είναι σαφές ότι επειδή δεν έχουν επιρροή στις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές, οι εθνικοί βουλευτές δεν τους ενδιαφέρουν, αλλά οι τοπικές βουλές και η τοπική αυτοδιοίκηση ε, ακούνε τώρα τη φωνή τους. Δεν είναι παραβίαση των δικαιωμάτων τους να τους αφαιρεθούν αυτά τα δικαιώματα. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακύρωσε ένα τμήμα του εκλογικού νόμου για τα άτομα ε, με προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν μπορούσαν βέβαια να ψηφίσουν παλιότερα όταν ήμουν ψυχίατρος, τώρα όμως μπορούν. Δεν είναι λοιπόν η απώλεια δικαιωμάτων ένα πρόβλημα. Γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια πολιτών της Ένωσης. Θα έπρεπε, αν έχουν ήδη εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, να παραμείνουν για να έχουν κάποια επιρροή στην πολιτική ζωή, έστω και περιορισμένη. Και για το πρόβλημα της ε, ακραίας κατάστασης για τα θέματα ασφάλειας. Αν όλα αυτά τα αναβάλουμε για τη δεύτερη φάση, μπορεί να μην υπάρξει καμία συμφωνία για το θέμα της Europol και του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Αν πρέπει να παραταθεί ομόφωνα η διαδικασία αποχώρησης, τι θα γίνει με την συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις ευρωεκλογέ του 19. Θα ήταν υποχρεωμένο να συμμετάσχει, να υπάρξουν υποψήφοι ή μπορεί αυτό να αποτραπεί με κάποιο τρόπο. Και για, τα απόλυτο, για το απόλυτο δικαίωμα Τη ελεύθερη διακίνηση, ε, πότε δεν ήταν απόλυτο το δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορία, ε, μπορεί να περιοριστεί για διάφορου λόγου, η δημόσια υγεία κτλ. Υπάρχει όμω μία ρύθμιση που λέει ότι μπορούν να υπάρξουν ε, όρια σε καταστάσεις έκτακτη ανάγκη, όπω στο Λίχτενστάιν. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να αξιοποιήσουμε αυτό για να θέσουμε ανώτατα όρια ε, στην ελεύθερη κυκλοφορία, να έχουμε μια συμφωνία τύπου Νορβηγίας και επειδή είμαστε ήδη στον ΕΟΧ, αυτομάτως θα φύγουμε όταν θα γίνει το Brexit στον ΕΟΧ ή θα πρέπει να ξαναμπεί στην ΕΖΕΣ και να υπογράψει την σύμβαση ΕΟΧ για να έχουμε μια λύση Νορβηγία συν Τελωνιακή Ένωση. Δεν υπάρχει σαφήνεια αν θα παραμείνει στον ΕΟΧ ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ή θα πρέπει να αποχωρήσει και να επανενταχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, δώσω το λόγο στην Diana James, θα ήθελα απλώ να σας πω ότι θα πρέπει να αποχωρήσω για να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή για ε, λίγο. Θα αναλάβει συνάδελφος την Προεδρία. Αλλά θα ήθελα ε, να σας αναφέρω κάποιες ε, ε ερωτήσεις που δημιουργούν κάποιες ανησυχίες. Παραδείγματος χάρη, τι δυνατότητα να σταματήσει ο χρόνος και επίση, ε, μία ερώτηση προ την καθηγήτρια Ντάγκλα Σκότ, διότι ήδη έγιναν πάρα πολλέ συζητήσει και στα πλαίσια της Σκοτία και ε, το γεγονός ότι ε, τα κοινοβούλια αυτά έχουν και κάποιες εξουσίες, όπως για παράδειγμα το Κοινοβούλιο της Σκοτίας, ε, ε, κάποιοι τομείς και πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι της αρμοδιότητάς τους. Επομένως υπάρχει δυνατότητα και λόγος να συμμετέχει το Σκοτικό Κοινοβούλιο για σχετικό νομοσχέδιο ε, κατάργησης ή ανάκλησης. Εσείς όμως είπατε ότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από πλευράς ε, Βρετανικής κυβέρνησης, ε, απλώς μόνο διαβούλευση. Δεν υπάρχει κάποια δεσμευτική ε, νομικά δυνατότητα διαβούλευσης. Μήπως θα μπορούσατε να μας τα εξηγήσετε και η γραμματεία θα σημειώσει ό,τι θα μας πείτε. Σας παρακαλώ μην θεωρήσετε λοιπόν ότι δεν ενδιαφέρομαι. Η Diane James. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο έθιξε ο κύριος Κόρμπετ, επομένω δεν θα τα πω εγώ. Ο κύριος ε, Τάγκον, ε, Τάνοκ ε, έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλιων, αναφέρθηκε στη λεγόμενη μεταβατική περίοδο και το τι θα έχουμε από άλλους ευρωβουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Επίτροπο και άλλους που έχουν υψηλά αξιώματα. Το τελευταίο μου σχόλιο, και εδώ απαντώ απευθείας στην κυρία Άντερσεν, διότι είχαμε διαφορές ε, στο παρελθόν, να ρωτήσω το εξή. Έστω ότι έχουμε μια σειρά από βουλευτέ ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στι ε, διαπραγματεύσει στο Brexit, αλλά δεν συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο του Westminster. Υπάρχει κάτι στο ευρωπαϊκό σύνταγμα, στο Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου που θα τους υποχρεώσει. Διότι αν είναι να δώσουμε φωνή σε κάθε ομάδα, σε όλα τα κράτη-μέλη, θα πρέπει λοιπόν να έχουν και αυτή την αναγνώρισή τους και να ακουστεί και η δική τους η φωνή. Αν θέλετε θα το απαντήσω αυτό, λέει η κυρία Άντερσεν. Ευχαριστώ και πάλι. Δεν έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, η κυρία Σκότ. Λοιπόν, για την ερώτηση για τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Με εκπλήσει το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει περισσότερη συζήτηση για το θέμα. Από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό που αναφέρεται είναι ότι η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει, σφέρει το πλαίσιο αλλά ε, δεν ε, ε, μπορεί να εκτελεστεί λόγω της συμμετοχής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια να συζητήσουμε, αλλά αν πρέπει να αναλάβει δράση κάποιος, η Ιρλανδία είναι αυτή η οποία θα πρέπει να δράσει και μέχρι τώρα η Ιρλανδία δεν έχει δείξει και μεγάλη διάθεση να δράσει. Ε, θα έλεγα ότι επαφίεται από αυτούς, σε αυτούς δεν περιμένω τίποτα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, για τους Ευρωπαίους πολίτες ε, και τα κεκτημένα δικαιώματά τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον πόσο μικρά είναι αυτά τα κεκτημένα δικαιώματα. Έκανα κάποια έρευνα πριν από ένα χρόνια και είδα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ε, πολύ λίγη προστασία που προσφέρεται στα κεκτημόνα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε και πριν ε, από την εκστρατεία για το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, δεν συζητούμε απλώς ε, Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολλούς ε, πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που χάνουν την ηθαγένειά τους. Και θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη δράση από νομική σκοπιά για να εφαρμοστούν αυτά. Είναι απογοητευτικό το γεγονό ότι δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο σε μεγάλο βαθμό. Αυτά που είπε η πρόεδρο για τη Σκοτία και την εκχώρηση εξουσιών προ αυτού. Ε, να πω το εξή. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των διαπραγματεύσεων ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συμφωνία Αποχώρησης που θεωρείται θέμα εξωτερικής πολιτικής, άρα εμπιστευτικό θέμα βάση του καταστατικού για την ε, ε, Σκοτία το 1998, γι' αυτό και δεν έχουμε και συμμετοχή του Σκοτικού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της Ιουαλίας και αν υπήρχε κοινοβούλιο και στη Βόρεια Ιρλανδία και αυτούς, και την ε, κατάσταση στο εσωτερικό. Όσον αφορά ε, το νόμο της ανάκλησης, το, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται ότι έχει αναγνωρίσει ότι θα υπάρξει ανάγκη για νομοθετική συγκατάθεση των κατατόπων κοινοβουλίων ε, διότι υπάρχουν θέματα που τους αφορούν ε, και είναι της αρμοδιότητάς τους. Γεωργία, αλία κλπ. που ε, έχουμε χωρίσει εξουσίες σε αυτά τα κοινοβούλια. Και αυτό διαφέρει από αυτό που λέει στη δεύτερη λευκή βίβλο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Λέει ότι δεν είναι απόλυτα σαφές πού θα πάνε αυτές οι αρμοδιότητες όταν θα επιστραφούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία ε, για την περίπτωση της Σκοτίας, ε, για παράδειγμα, λέει ότι εκχωρούνται πλήρως, σαφέστατα αυτές οι εξουσίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι θα συμβεί εάν ε, τους αρνηθούν αυτές τις εξουσίες. Αυτό θα οδηγήσει σε συνταγματική κρίση. Σίγουρα λοιπόν είναι ένα από τα πολύ σημαντικά σημεία για την εσωτερική διαδικασία του Brexit. Τέλος, την παρατήρηση της Diane James, η οποία νομίζω ότι αποχώρησε. Αν μπορούν ε, να υποχρέωσουμε κάποιους βουλευτές να αναλάβουν ε, την έδρα τους. Ε, το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα ήθελε να παρέμβει σε καμία περίπτωση με το Εθνικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Συγγνώμη, διορθώνω η ομιλήτρια. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα παρέμβει στο εθνικό συνταγματικό δίκαιο. Γι' αυτό είχαμε και την υπόθεση Μίλλερ στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δούμε ε, ποιε είναι οι συνταγματικές απαιτήσει για την ενεργοποίηση του άρθρου 50 ευθύ εξ αρχή. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι θα ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό. Η κυρία Άντερσεν χωρίς μικρόφωνο σχολιάζει. Ο κύριος Σέκχαλτ, καθηγητής Σέκχαλτ. Για πρώτερη, αρχική συμφωνία για δικαίωμα των πολιτών και ότι τίποτα να έχει συμφωνηθεί, μέχρι συμφωνηθούν τα πάντα. Από πλευράς νομοθεσίας δεν μπορώ να δω γιατί να μην μπορεί να υπάρξει ένα σχέδιο αρχικό συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών και προσωρινά να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία μέσω εσωτερική εφαρμογής στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, είναι δυνατόν να εφαρμόσετε προσωρινά μια συμφωνία πριν να συναυθεί τελικά. Κανονικά βέβαια πρέπει να υπάρχει πλήρη συμφωνία και να εφαρμόσετε αυτή προσωρινά. Δεν βλέπω να υπάρχει νομικό εμπόδιο να συναυθεί μια συμφωνία για αυτά τα δικαιώματα και να αρχίσει η εφαρμογή αυτής. Εν αναμονή των, της ολοκληρώσεως των διαπραγματεύσεων. Μία ενιαία συμφωνία με διπλή νομική βάση και έγκριση κρατών μελών. Εάν θα συνεπάγεται έγκριση των κρατών μελών. Εξαρτάται. Σε πραγματικούς όρους στην πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής Ενώσης είναι εφικτό. να η νομοθεσία να χρησιμοποιήσει τη νομική βάση για τη, τη συνθήκη τη λειτουργία Ευρωπαϊκή Ενώσεω για τη σύναψη συμφωνία σύνδεση, οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι πολύ ευρείε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι μια σύνδεση συνεπάγεται συμμετοχή σε οποιαδήποτε πολιτική έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνδεδεμένη χώρα που συμμετέχει και είναι δυνατόν νομικά να υπάρχει συμφωνία σύνδεσης με πολύ ευρύ φάσμα που συνάπτει μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρακτικά όμως είναι μεικτέ αυτές οι συμφωνίες σύνδεσης. Από πλευρά νομική όμω δεν απαιτείται κάτι τέτοιο. Ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τι με τις γνώμες του, πάντα με ενοχλούσε αυτό, αλλά σε κάποιε περιπτώσεις ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου για κάποια επικείμενη συμφωνία, αλλά οι θεσμοί προχώρησαν με τη σύναψη και το δικαστήριο είπε ότι δεν είναι αποδεκτή μια γνωμοδότηση διότι υπάρχει ενδεχόμενη συμφωνίας. Δεν ξέρω τα μέρη της συμφωνίας πρέπει να επιτρέψουν στο, στο δικαστήριο να το, τοποθετηθεί πριν συνάψουν τη συμφωνία. Και η διετής περίοδος Ποια είναι. Το άρθρο 50 λέει ότι η διετής περίοδος είναι περίοδος αποκοπής που εφαρμόζεται μόνο όταν είναι σαφές ότι δεν υπάρχει συμφωνία, καμία συμφωνία, διότι λέει αποτυχώντος αυτού, αποτυχούσης της συμφωνίας, αν υπάρχει μια συμφωνία που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης που δεν έχει τεθεί σε ισχύ, διότι πρέπει να εγκριθεί από όλα τα μέρη, τότε εκεί πρέπει να αναστέλλεται ο χρόνος για τη διετή περίοδο. Αλλιώς έχουμε το αποτέλεσμα του άρθρου 50 που είναι ένα φαινόμενο γιλοτίνας, αποκόπτη. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ούτω ώστε το κράτο μέλο πάντα που θέλει να αποχωρήσει να μπορεί να αποχωρήσει ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία. Αν όμω υπάρχει συμφωνία που είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεω, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συμφωνώ, υπάρχει ένα κίνδυνο μιας του διαζυγίου αυτού με ελάχιστη κάλυψη και θα είναι αρκετά περιορισμένη η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων ενδεχομένω και η συμφωνία αυτών όσον αφορά μια περιορισμένη εμβέλεια διευθέτηση. Και πραγματικά υπάρχει πρόβλημα δημοκρατικής φύσης και εκτιμένα δικαιώματα. Και το δικαίωμα ψηφοφορίας στις δημοτικές εκλογές και αν αυτό αποτελεί παραβίαση μελιωδών δικαιωμάτων. Δύσκολο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επιχειρηματολογήσει κανείς. Δεν το έχω εξετάσει το θέμα εις βάθος όμως. Ε, ε, εάν η απώλεια δικαιώματος ψηφοφορία σαν αποτέλεσμα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτό απαραίτητα αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξετάσαμε κάπως το θέμα των κεκτημένων δικαιωμάτων και πώς έχει διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ έχουμε μοναδική περίπτωση. Δύσκολο να εξετάσουμε προηγούμενο. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Κάποιοι να έχουν χτίσει τη ζωή τους πηγαίνοντας να κατασταθούν σε άλλο κάτω μέλος και μετά από 20-30 χρόνια να αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι αυτή η χώρα αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα δικαιώματά τους χάνονται. Κατά την άποψή μας υπάρχουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τίθεται με ένα μοντέλο Brexit ή εξόδου που σημαίνει το δικαίωμα απασχόλησης, τα δικαίωματα αποφυγής διακρίσεων, τα δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης, όλα αυτά χάνονται ξαφνικά. Και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το ΔΕΚ θα αποφασίσουν πιθανότατα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου αν παραταθεί η περίοδος αχορτογράφητη η περιοχή αυτή. Είδαμε πάρα πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την πάροδο των ετών σε δύσκολες κρίσεις και πολιτικές περιστάσεις που θα μπορούσαν να εξεταστούν ο πλευράς καθαρής εφαρμογής του νόμου. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να παρατείνει την περίοδο των διαπραγματεύσεων και να αποφασίσει ότι δεν θα δεξαχθούν εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις επόμενες ευρωεκλογέ. Διότι, εν πάση περιπτώσει, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αν αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής, δεν ξέρω, έχουμε δει και χειρότερα, χειρότερες αποφάσεις από αυτήν που έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτόματη αποχώρηση από την Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Υπάρχουν κάποια ακαδημαϊκοί που διατείνονται ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποσυρθεί από τον ΕΟΧ ρητά, παραμένει μέρος αυτού, εγώ δεν έχω πιστεί. Υπάρχει όμως ένα γενικό πρόβλημα με άλλες πολλές διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μπορούν να συνεχίσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν δεν θα είναι πλέον κάτω μέλος, αλλά επίσης απαιτούν μία απόφαση απόσυρσης ή επαναδιαπραγμάτευσης. Και όλα αυτά αποτελούν ένα κομμάτι του θεματολογίου του Brexit. Το ερώτημα της κυρίας Προέδρου για το να σταματήσουμε το χρονόμετρο αναφέρεστε κυρίως στη δυνατότητα ανάκλησης της κοινοποίησης του άρθρου 50 της, ένα του άρθρου 50. προσωπική μου άποψη και η πλειοψηφία των ειδικών για την ευρωπαϊκή νομοθεσία όχι όλων, της πλειοψηφία. Αν ληφθεί μια σοβαρή απόφαση σε επανεξετάσεω, όχι απόφαση που λέει ότι σταματάμε το χρονόμετρο και σε ένα χρόνο ξαναρχίζουμε και πάλι, αν ληφθεί μια σοβαρή απόφαση επανεξέτασης και ριζικής αναστροφής της αποφάσεως εξόδου την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 50 παράγραφος 1, ένα κάτω μέλος δύναται να αποφασίσει, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά θα υποχρεωθεί να αποχωρήσει το κράτος μέλος. Η έννοια ποια είναι του, κράτου, του άρθρου 50. Το δικαίωμα του κράτους μέλους σύμφωνα με τα συνταγματικά του δικαιώματα μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει ένα κράτος μέλος αντικατοπτρίζει το σεβασμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο και τους συνταγματικούς κανόνες σε εσωτερικό επίπεδο. Αν γίνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα ή κάποια πράξη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία σταματά το Brexit, τότε θα σταματήσει το ρολόι. Θα πρέπει να πετάξουμε το ρολόι, βασικά, το παράθυρο. Για το ανασταλικό αποτέλεσμα της απόφασης. Θα έπρεπε να μπει μια ρήτρα στην ίδια τη συμφωνία που θα έλεγε ότι εάν τυχόν ζητηθεί γνώμη του δικαστηρίου για τη συμβατότητα με τις συνθήκες θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. για τα δικαιώματα των πολιτών. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να γίνουν ε, μονομερείς δηλώσει και των δύο πλευρών ή μία ανταλλαγή επιστολών. αυτό που λέτε για το ότι θα μπορούσε να ισχύσει το status quo για μια σειρά ετών, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο επιθυμητή μετάβαση. Οι καθευτήρες γραμμές αναφέρουν διάφορες αρχές. Ακεραιότητα της ε, νομικής τάξης της Ένωσης, ε, αυτομία των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μπορεί να υπάρξουν πολλά προβλήματα αν ε, η μεταβατική περίοδος δεν σημαίνει πλήρης εφαρμογή του κοινωτικού κεκτημένου και δυνατότητα δικαστικού ελέγχου. Αλλά εφόσον είναι μεταβατική περίοδος, μια περίοδος δηλαδή που θα αρχίσει να ισχύει μετά την ε, τυπική αποχώρηση, τότε θα, δει, το θέμα των συμμετοχικών δικαιωμάτων. Σε μια μεταβατική περίοδο θα είχε δικαίωμα συμμετοχή στον Ηνωμένο Βασίλειο. Βασίλειο. Εγώ νομίζω ότι δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως μια υποψήφια χώρα που έχουν υπογράψει τη συνθήκη ένταξη θα έπρεπε να έχει ένα καθεστώ παρατηρητή στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο κτλ. και την Επιτροπή. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ίσως μια διαφοροποιημένη ρύθμιση. Το να έχουν ένα δικαστή και έναν ε, εισαγγελέα θα μπορούσε να βοηθήσει για να νομιμοποιείται αυτή η ρύθμιση για την διπλή νομική βάση. Συμφωνώ με αυτά που λέει ο Πίτα. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο άρθρο 50, μια συμφωνία άρθρου 50 και μια συμφωνία σύνδεσης. Η συμφωνία σύνδεσης απαιτεί ομοφωνία, άρα θα επανέρχεται, θα, θα επανέρχεται το βέτο. Θα πρέπει να είναι χωριστέ λοιπόν αυτές οι δύο νομικές βάσεις, γιατί είναι ασύμβατες. Η αναφορά στο 3, 5 και το 8 ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι τμήμα του συνταγματικού πλαισίου εντό του οποίου λειτουργούν οι διαπραγματευτέ. Είναι μόνο ένα παράδειγμα για το τι πρέπει να έχουν κατά νου κατά τη διαπραγμάτευση. Το άρθρο 8 Βεβαίω είναι σημαντικό για τη στιγμή που θα αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει γειτονικό κράτος με το οποίο δεσμεύεται μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας η Ένωση να έχει ειδικέ σχέσεις με συγκεκριμένους στόχους. Άρα τα άρθρα αυτά που αναφέρονται στο προήμιο του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικά για το πώς θα γίνουν πραγματεύσεις και για την ένταξη και για μια μελλοντική συμφωνία. Αν ε, μείνει περισσότερο το Ηνωμένο Βασίλειο, θα έπρεπε να έχει ευρωβουλευτέ. Αυτό εξαρτάται από το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Για παράδειγμα, είπε ότι δεν θέλει να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι δεν προτίθεται πλέον να αναλάβει την Προεδρία. Θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να πει, κοιτάξτε, εντάξει, μένουμε. Αλλά δεν θα οργανώσουμε τώρα, διοργανώσουμε προεκλογέ. Και ποιο θα συμμετάσχει σε μια προεκλογική εκστρατεία. Ποιο θα είναι υποψήφιο για ένα χρόνο στο Κοινοβούλιο και μετά, άντε για. Αλλά αν θέλει να το κάνει, α το κάνει. Εφόσον παραμείνει για μερικά χρόνια ακόμη επειδή, επειδή θα παραταθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης, βεβαίως είναι κράτος μέλος. Θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να διοργανώσει ευρωεκλογέ. Ίσως και την υποχρέωση. Και τότε γιατί δεν είχε υποχρέωση να λάβει και την Προεδρία. Τάνοκ. Ναι, αν παραμείνει παρά παρατείνει συγγνώμη, για πάνω από λίγους μήνες, ε, τότε θα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει εκλογές. Και, γιατί τότε δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν τα 3 εκατομμύρια πολίτε και δεν θα έχει εκπροσώπηση για την νομοθεσία. Αλλά και τι θα κάνουν οι υποψήφοι. Μα πάντα μπορεί να βρει υποψήφιου, λέει ο κ. Στάνο. Τώρα, για την αποχώρηση από τις συμφωνίες ε, ΕΟΧ. Η γραμματεία του ΕΖΕΣ έχει από πλευράς νομικών εμπειρογνωμόνων την άποψη ότι όταν θα αποχωρήσει από την Ένωση πάβει να ανήκει στον ΕΟΧ γιατί δεν θα ισχύει πλέον το 126 για την ε, γεωγραφική έκταση εφαρμογής. Εφόσον δεν θα είναι πλέον μέλος της Ένωσης, εξορισμού δεν θα εφαρμόζεται στον Ηνωμένο Συμφωνία ΕΟΧ. η νομική υπηρεσία του Νορβηγικού Υπουργείου Εξωτερικών έχει την ίδια άποψη. Και νομίζω ότι την ίδια άποψη έχει και η Βρετανική μόνιμη αντιπροσωπεία. Αλλά ίσως χρειάζεται κοινοποίηση για να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν ενδιαφέρεστε, μόλις έκανα, ολοκληρώσα μία έκθεση για την ορική κυβέρνηση για τις επιπτώσεις ε, στον ΕΟΧ του Brexit. Υπό ποιε συνθήκε θα μπορούσε να σταματήσει το ρολόι. Νομίζω πως ήταν δύσκολο για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να πετάξει με τις κλωτσιές ένα κράτος μέλος που εξακολουθεί να είναι κράτος μέλος. Δεν υπάρχει νομική βάση γι' αυτό. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Ένωση είναι να αναστείλει κάποια από τα δικαιώματα που απορρένουν από την Ένωση. Και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό από τη συμμετοχή στην Ένωση. Αλλά αν υπάρχει μια σοβαρή δημοκρατική απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μείνει τελικά στην Ένωση, τότε η Ένωση δεν έχει άλλη δυνατότητα από το να πει καλά εντάξει. Αλλά δεν νομίζω ότι από μόνο του το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία. Θα πρέπει κάπως ε, να είναι απόρρεα διαπραγματεύσεων. Το άρθρο 50 δεν λέει τίποτα. Είναι ασαφές. Αλλά επειδή μόνο στην παράγραφο 1 γίνεται αναφορά στην εσωτερική διάσταση της ε, απόφασης αποχώρησης, η διαδικασία στη συνέχεια γίνεται με συμμετοχή των θεσμών. Άρα δεν μπορεί από μόνο του το Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει τη διαδικασία. Και αν ήμουν μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τότε θα ήθελα πολύ σοβαρές διαβεβαιώσεις ότι δεν σταματάνε για να ξαναρχίσουν τη διαδικασία αποχώρηση μετά από κάνα δύο χρόνια. Αλλά υπάρχει και άλλη άποψη. Υπάρχει και η τελευταία παράγραφος που λέει ότι το άρθρο 49 εξακολουθεί να ισχύει και, να μπορεί, και μπορεί να αξιοποιηθεί. Οπότε το θέμα κυρίως είναι σε ποια στιγμή τη διαδικασία το θέμα της ε, ακύρωση τίθεται. αν είμαστε κοντά στο τέλος. Και ακόμη αν το Κοινοβούλιο απορρίψει τη συμφωνία λέγοντας ότι θα προτιμούσε την παραμονή του ΕΒ δεν νομίζω ότι θα αρκούσε για να πιστούν όλα τα κράτη-μέλη ότι είναι επαρκέ αυτό για να σταματήσει η διαδικασία και να επανέλθουμε στο status quo ante. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία πολύ σύντομη ερώτηση προς τον καθηγητή Eichhout για τη δυνατότητα ανάκληση του revocability. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι το δημοψήφισμα για το Brexit θα μπορούσε να ανακληθεί μέσω άλλου δημοψηφίσματος ή μέσω απόφασης του Κοινοβουλίου. Πιστεύετε ότι συνταγματικά υπάρχει το ενδεχόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, νομίζω ότι η απόφαση Μίλλερ το καθορίζει αυτό, διότι και το Ανώτατο Δικαστήριο και ο Άριος Πάγος ουσιαστικά είπαν ότι το δημοψήφισμα ήταν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και χρειαζόταν ψήφος του Κοινοβουλίου για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πλευρά σταγματικού δικαίου λοιπόν το Κοινοβούλιο αρκεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, για να ε, συζητήσουμε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να ζητήσω και από τους τρεις σας, εξ ονόματος της Προέδρου, ή δυνατόν να μας στείλετε τις ομιλίες σας στη γραμματεία και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Η υπηρεσία PRS μας ε, ενημέρωσε ότι υπήρχε, υπάρχει μια πρόσφατη δημοσίευση για την αναχώρηση, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αναφέρει και αρκετούς ε, από τους γράφοντες. Έχουμε τα σχετικά έγγραφα εδώ στην αίθουσα αν σας ενδιαφέρουν. Και η γραμματεία θα συμπεριλάβει και την, ε, το σύνδεσμο αυτού του εγγράφου στην ιστοσελίδα που αφορά το Brexit. Ε, I, would like to ask Mr. Corbett. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Κόρμπετ να μας παρουσιάσει τα της ερμηνείας του άρθρου 5 και 210α του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι άλλαξε νωρίτερα η διάταξη για να ακούσουμε τώρα την έκθεση του κυρίου Πρέντα, αλλά έχω ένα πρόβλημα, πρέπει να φύγω για άλλη συνεδρίαση. Ο κύριο Βίλαντ βέβαια δεν έχει έρθει ακόμα. Θα σα παρουσιάσω εγώ λοιπόν τα πράγματα στα γρήγορα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τεχνικό και ε, αρκετά δύσκολο. Ερμηνεία λοιπόν των άρθρων 5 και 210α του κανονισμού. Πρόκειται για ένα τεχνικό ξεκαθάρισμα λόγω των μεγάλων αλλαγών που κάναμε στον κανονισμό το Δεκέμβριο, αλλά υπάρχει ένα σημείο στο οποίο δεν ήταν αρκετά σαφής ο κανονισμός για το για την ιεράρχηση των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια ιεράρχηση. Οι συνθήκες είναι οι πιο σημαντικές, η νομοθεσία θα πρέπει να συνάδει με τις συνθήκες, οποιαδήποτε διοργανική συμφωνία θα πρέπει να συμμορφούνται με την νομοθεσία και με τις συνθήκες και ε, ο κανονισμός ενός ε, θεσμικού οργάνου θα πρέπει να συμμορφούνται με όλα τα παραπάνω. Επομένως, εδώ απλώς προσθέτουμε μια ερμηνεία για να διευκρινίσουμε ότι όντως συμβαίνει αυτό και έχουμε και την σωστή υποσημείωση ε, που παραπέμπει στη Συμφωνία Πλαίσιο που πρόκειται για διοργανική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γίνονται απλώ αυτά για λόγου διευκρίνηση, δεν προστίθεται κάτι παραπάνω, δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Merci euh, infiniment, Président. Χίλια ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ξεκινάω βέβαια αν με σταματήσει ο, σόρ, θόρυβος γιατί είναι ε, εκνευριστικός. Σας παρακαλώ πολύ. Χίλια ευχαριστώ και πάλι. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα, για την ηθαγένεια και χαίρομαι που η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων μπορεί να γνωμοδοτήσει για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η ηθαγένεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση από τότε που εισήχθη αυτή η έννοια στη συνθήκη του Μάστριχτ. Ε, κάποια στοιχεία λειτουργούν αποτελεσματικά και νομίζω ότι θα πρέπει να χαιρόμαστε που ε, σε αυτή την περίοδο που σοβεί ο λαϊκισμός μπορούμε να βάλουμε στην άκρη ε, τα ε, κεκτημένα και να επικεντρωθούμε στα αρνητικά. Λες και υπάρχουν αρνητικά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε πολλά στην Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια με καλά αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Παραδείγματο χάρη να ταξιδέψουν, να σπουδάσουν, να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα υπάρχουν βελτιώσεις, ε, ε, για παράδειγμα συμμετοχή στις ευρωεκλογές το ενδιαφέρον των πολιτών για τις ευρωεκλογέ ε, και το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρονται είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Η συμμετοχή μειώνεται σταδιακά σε κάθε νέα εκλογική αναμέτρηση ε, και στις ε, πρόσφατες ε, αλλαγές που κάναμε πάλι δεν βελτιώθηκε η συμμετοχή. Και πρέπει φυσικά να συνειδητοποιήσουμε ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε μια σωστή λύση. Στη γνωμοδότηση αυτή προσπάθησα να σταθώ σε κάποια σημεία γιατί ήταν και σύντομη. Έχω την εντύπωση ότι πιο πολύ μίλησα παρά έγραψα τη γνωμοδότηση, τη γνωμοδότηση, αλλά αυτά είναι τα όρια τα οποία επιβάλλονται βάσει διαδικασίας. Θα σταθώ λοιπόν καταρχάς στο θέμα της ε, μεταρρύθμισης ε, του εκλογικού νόμου, πρέπει οι ευρωεκλογέ να γίνουν πιο πολιτικού χαρακτήρα για να μπορέσουν να ε, έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών. Χρειαζόμαστε βεβαίως περισσότερη ε, διαφάνεια. Αυτό βέβαια ξέρω ότι εκνευρίζει πολύ συχνά τους πολίτες, να ενημερώνουμε περισσότερο τους πολίτες και εγώ προσωπικά φρονώ και νομίζω ότι έχει γίνει ήδη και σχετική μάχη εδώ, πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την ηλεκτρονική ψήφο. Δεν είχε αποτέλεσμα, δεν τα καταφέραμε καν εδώ στην Επιτροπή μας να έχουμε πλειοψηφία, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο συζητιέται όλο και περισσότερο και ε, προσφέρει περισσότερα στον καθένα. Κάνουμε τόσα πολλά πράγματα μέσω της ηλεκτρονικής οδού, γιατί να μην μπορεί να γίνει και αυτό, ε, λοιπόν, να μην ψηφίσουμε και ε, ηλεκτρονικά. Και επίσης πιστεύω ότι το θέμα του Brexit είναι θέμα ε, μείζωνος ανησυχίας για τους Ευρωπαίους πολίτες και το διαπιστώνουμε και από τον αριθμό των αναφορών που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Αναφορών θα τη συζητήσει αυτέ τι αναφορέ αύριο. Έχω πάρα πολλά αύριο να κάνω στην Επιτροπή Αναφορών για τι αναφορέ αυτέ που αφορούν το Brexit και είναι από όλε τι χώρε. Αφορούν θέματα που θα, θα μπορούσε κανείς να φανταστεί έτσι ευθόρμητα. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να θέσουμε μια απλή προτεραιότητα, να θέσουμε στο επίκεντρο τον, τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών, να υπάρχει αυτό η συμφωνία, να δούμε την ασφάλεια δικαίου και να επιμείνουμε για την ελεύθερη κυκλοφορία και την ελεύθερη διαμονή και δικαίωμα ψήφου για τους ανθρώπους που διαμένουν σε μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτά λοιπόν ε, ε, είναι το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να θίξω στη γνωμοδότηση και ένα τρίτο που θεωρώ εξίσου σημαντικό η ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Η ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βελτίωσης της νομοθεσίας ε, μέσω τροποποίησης της είναι κάτι πάρα πολύ καλό και δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή την πρωτοβουλία. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τη χρήση και να επιτρέψουμε στους Ευρωπαίους πολίτες που δεσμεύονται για κάποιο θέμα να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο και να μην απομακρύνονται για την πολύ περίπλοκη διαδικασία. Ε, μπορεί να επιτύχουμε τελείω διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε. Επίσης, θέλησα να επισημάνω τις προσπάθειες που έγιναν σε θέματα ασφάλειας. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω που θίγει και η γνωμοδότηση. Η ασφάλεια ε, είναι θέμα που ανησυχεί τους πολίτες μας και επομένως αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα κάθε φορά που μιλάμε για ηθαγένεια. Η ασφάλεια είναι ζωτική σημασία, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε περαιτέρω μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρχει ε, περισσότερη ασφάλεια και παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια είναι αρμοδιότητα κυρίως των κρατών μελών, έχει ρόλο να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν με λίγα λόγια περιλαμβάνονται σε αυτή την πολύ σύντομη γνωμοδότηση. 1500 χαρακτήρες όλοι και όλοι. Ε, τηλεγράφημα στέλναμε παλιά, δεν έχουμε πια τηλεγραφήμα, αλλά τέτοιο είναι. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ κυρία Πέντα Κυρία Παπαρδέν και στους άλλους κοιόδης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Τον ευχαριστώ που ετοίμασε αυτή τη γνωμοδότηση του ΕΛΚ. Θα ήθελα να εξηγήσω ποια είναι η δική μου θέση που εκφράζεται μέσω τροπολογιών. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και πολύ. Διάβασα την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έγιναν δημόσιες διαβουλεύσεις και δημοσκοπήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει τέσσερα βασικά στοιχεία για το θέμα αυτό. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Θέλω να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές που θεωρώ σημαντικές. Πρώτον, ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν το καθεστώς τους, ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πολλοί που θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους και ο αριθμός τους αυξάνεται. Αυτό πρέπει να μας ικανοποιεί. Είναι κάτι που μας ενθαρρύνει να εργαστούμε περισσότερο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεύτερον, 4-5 Ευρωπαίους εκτιμούν την ελευθερία μετακίνησής τους, που μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν σε μια άλλη χώρα και να ασκούν και εμπορικέ δραστηριότητες σε άλλες χώρες. Αυτές οι θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι δικαιώματα από τα οποία δεν θέλουμε να παρετηθούμε. Γι' αυτό και στις διαπραγματεύσεις για το Brexit πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνέχιση ισχύω των κεκτημένων δικαιωμάτων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και που έχουν ωφεληθεί από την ελευθερία μετακίνησης. Πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είπαν ότι δεν είναι απόλυτα σίγουροι για τα, νομικά τους, για νόμιμά τους δικαιώματα και δεν ξέρουν σε ποιο να στραφούν όταν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους ή όταν υπάρχει κάποια παράβαση. Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους πιστεύει, πιστεύουν ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές αν ο κόσμος είχε περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή του. Θα ήταν χρήσιμο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν περισσότερα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των πολιτών, διότι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι το παρόν επίπεδο πληροφόρησης είναι ανεπαρκές. Κατά την άποψή μου, η ανταλλαγή απόψεων και οι συζητήσεις με τους πολίτες είναι ένας τρόπος βελτιώσεως της ευαισθητοποίησης του λαού ε, για τον αντίκτυπο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Οι εθνικές και τοπικές αρχές έχουν ρόλο να διαδραματίσουν και θα πρέπει να μπορούμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους σε σημαντικό βαθμό. Περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι τα τρία επίπεδα συνεργασίας που θα πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω. Τέλος, εξίσου σημαντικό, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του, να γνωρίζει ότι μπορεί να απολαμβάνει αυτά τα δικαιώματα όταν εργάζεται, ζει και ψηφίζει και να μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του στον τόπο διαμονής του. Στην έκθεση του 2017 μάλλον μετά την έκθεση του 2017 και κατά τη διάρκεια του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει εκστρατείε ευαισθητοποίησεω σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, δικαιώματα παροχή αρρωγή από τι πρεσβείε, δικαιώματα ψήφου κλπ. Ο κ. Πρέντα αναφέρθηκε στι στοιχέ τη ασφάλεια. Και αυτό το θέμα από μόνο του γίνεται ένα δικαίωμα και είναι ζωτική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν τρόπο αυτό το δικαίωμα να το υλοποιήσει, να το μεταφράσει σε πραγματικότητα. Χρειάζεται περισσότερος συντονισμός μεταξύ μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτός είναι ένας τρόπος καταπολεμήσεως της τρομοκρατίας και προστασίας των πολιτών μας. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα και υπάρχει προσδοκία πλευράς των πολιτών της Ευρώπης να αντιμετωπιστεί. 2018-2019 Εκεί στόχος θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάρμπαρα Σπινέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ τον συνάδελφο τον κύριο Πρέντα και ελπίζω ότι θα κατορθώσουμε να συνεργαστούμε με τον πιο καρποφόρο τρόπο. Πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο μέσω πολλαπλών εκθέσεων και μέσω αυτού του κειμένου που είναι μια γνωμοδότηση θα ήταν σκόπιμο να δώσουμε μια απάντηση σε δυσαρέσκεια των πολιτών, υφίσταται αυτή η δυσαρέσκεια και αυτή εκφράζεται μέσω υψηλών ποσοστών αποχής, εκφράζεται μέσω κινημάτων κατά της διαφθοράς, εκφράζεται και μια έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις πολιτικές, τις τάξεις των πολιτικών και των διαφόρων κυβερνήσεων. Πάνω σε αυτό μπορούμε να εργαστούμε, είμαι πολύ ικανοποιημένη που ο συνάδελφος Πρέντα αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες των πολιτών, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τίνει να μην το αναφέρει αυτό συχνά, αντιθέτως εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το κείμενο είναι αναγκαίο να είναι σύντομο, αλλά σε αυτό το πολύ σύντομο κείμενο θα ήθελα να υπάρχει και μια αναφορά στη σημασία να δοθεί υπόσταση στον κοινωνικό πυλώνα να αναφέρεται στην ηλεκτρονική δημοκρατία ή e democracy, το αναφέρατε ήδη. Και αυτό να είναι ένα συμπλήρωμα των παραδοσιακών μέσων ψηφοφορίας και πολιτικής συμμετοχής θα μου άρεσε, θα με ικανοποιούσε να υπενθυμίζει το δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή όταν τίθεται θέμα ελήψεως διαφανίας και κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρεται. Ο μηχανισμός Ίντφελτ για το έλεγχο της ισχύω του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όχι μόνο στα κράτη-μέλη, αλλά και μεταξύ θεσμικών οργάνων. Αναφέρεται αυτό στο μηχανισμό Ίντφελτ. Δεν αναφέρεται συχνά, αλλά είναι σημαντικότατος μηχανισμός που υπερψήφισε το Κοινοβούλιο. Και τέλος, δεν θέλω να έχω ένα μοκροσκελέστατο κείμενο, αλλά το τελευταίο που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου είναι ο δημοκρατικός έλεγχος της νομοθετικής διαδικασίας. Να γίνεται μια αξιολόγηση συνεπιών, impact assessment, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι υποχρεωτική αυτή η αξιολόγηση όταν θεσπίζεται νομοθεσία. Θα δώσει αυτό μια καλή εντύπωση, καλή εικόνα στους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις. Δεν ξέρω αν Ντάν να πεις τίποτα. Σημείωσα. Θα σας αποστείλω το κείμενο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα από αυτού. Ευχαριστώ. Έχουμε την συνάντησή μας στις 12 Ιουλίου όπου θα συζητήσουμε το σχέδιο νομοδότησης, θα θέσουμε την προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Μάλλον θα είναι 6 Σεπτεμβρίου, άρα θα υπάρξει κάποιος χρόνος. Ωραία. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό και περνάμε σε αυτά τα οποία περάσαμε, δηλαδή τα πηδήξαμε. η ερμηνεία των κανόνων 5 και 210 ο κύριος Κόρμπιτ ξεκίνησε τη συζήτηση να δώσω το λόγο στον κύριο Βίλαντ Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι Πρόκειται για μια σύγκρουση μεταξύ κάποιων συμφωνιών και του ιστορικού μας κανονισμού. Υπήρξε μια ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του κανονισμού, η οποία διαπίστωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αντίφαση μεταξύ της διατύπωσης ε, του κανονισμού και των ε, διαθεσμικών οργάνων του 10 και του 14 για την ε, χρήση εμπιστευτικών εγγράφων. Η προτινόμενη ερμηνεία βασίζεται σε αυτές τις δύο συμφωνίες και λέει ότι πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν αυτές οι δύο συμφωνίες. Συμφωνούμε με μία βράχη πρόθεσμη ερμηνεία γιατί πρέπει να αντιδράσουμε σύντομα αλλά σε κάθε περίπτωση τα άρθρα αυτά 5 και 210α όπως ε, ε, λέει και ο κύριος Γεραντόφσκι που ασχολείται με αυτό το θέμα, θα πρέπει αυτά τα άρθρα να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση του κανονισμού. Εξετάσαμε το θέμα αυτό, αλλά ορισμένα μας διέφυγαν. Πρέπει λοιπόν να τα ξαναδούμε αυτά. Και συμφωνήσαμε στη σχετική ομάδα εργασίας ότι δεν θέλουμε να έχουμε πολλές ερμηνείες. Καλύτερα να υπάρχουν σαφή κείμενα. Αλλά τελικά συμφωνώ να συμπεριλάβουμε κάποιες ερμηνείες στο κείμενο και κατόπιν όταν θα κάνουμε αποτίμηση και όχι αναθεώρηση θα έλεγα της όλης προσπάθειας να δούμε πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στο κείμενο. Η περαιτέρω επεξεργασία αυτών των ε, άρθρων θα συνδέονται και με το δικαίωμα δημιουργίας ειδικών επιτροπών έρευνας του Κοινοβουλίου. Συμφωνεί ο κύριος Κόρμπετ, έχετε τα κείμενα. Ο 5, το άρθρο 5 ιδιαίτερα η παράγραφος 5 μας ενδιαφέρει. Έχετε και το 210α, όπου κυρίως μας ενδιαφέρουν οι παράγραφοι 3 και 4. Και θα σας υποβάλω, αλλά μόνο στα αγγλικά, ένα κείμενο ερμηνείας. Δεν είναι και κοσμιστορικά αυτά τα θέματα. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Ούτως ώστε να τα αναγγείλουμε στην επόμενη ολομέλεια και να τα συμπεριλάβουμε ως ερμηνείες των σχετικών παραγράφων στο κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Θέλει η Επιτροπή να πάρει το λόγο. Όχι. Καλά. Α, δεν υπάρχει κανείς για αυτή την έκθεση. Α, ρωτάω γιατί δεν ξέρω.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 Are you Yeah. Λοιπόν, το έχετε λάβει. Το έχετε λάβει. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε. Είστε σύμφωνοι. Ξέρουμε επί ψηφίζουμε. Το κείμενο το έχετε. Λοιπόν, να ψηφίσουμε διανατάσεως. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ αυτών των νέων ερμηνεών όπως αναφέρεται στο κείμενο το αρχικό. Κατά παρακαλώ. Αποχές. Ωραία. Πανψηφί. Οπότε έκλεισε αυτό το θέμα. Συγγνώμη. Μήπω θέλει να μιλήσει για την έκθεση Πρέντα κανεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να ρωτήσω, αλλά όχι κανεί, όχι καλά, εντάξει. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα της μέρης της διάθεσης που είναι ο Γενικός Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 όλα τα τμήματα η Επιτροπή υπέβαλε την κατάσταση προβλέψεων για τον προβλησμό του 18 στις 29 Μαΐου 17 σας παρακαλώ όσοι θέλουν να, συζητούν, να βγουν σε αυτή την κατάσταση προβλέψεων από την Επιτροπή βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια μείωση για την Ευρώπη των πολιτών μια μικρή αύξηση για τα δικαιώματα, την ισότητα και την υπηκότητα Γι' αυτό προτείνω μέσω του σχεδίου γνωμοδότησης να εγκρίνουμε το κείμενο της Επιτροπής και όταν θα χρειαστεί να αντιτεθούμε σε ιεσδήποτε περικοπές από το Συμβούλιο. Για το 2018 η επικοινωνική μας πολιτική είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες λόγω των επικειμένων εκλογών του 19. Το δεύτερο στοιχείο θα θυμάστε ότι ως ΑΦΚΟ προτείναμε κάποιες προπαρασκευαστικές και πιλωτικές δράσεις, τέσσερις όλες μαζί. Είναι στη φάση της προκαταρκτικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε μέχρι τέλος Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί για να έχουμε χρόνο για να γίνει τελική ψηφοφορία στην ψηφοφορία μας, στην ε, συνεδρίασή μας τον Ιούλιο. Ξέρετε ότι για τις τροπολογίες του προπολογισμού είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος Δεν έχουμε φυσικά συνεδρίαση τον Αύγουστο, η πρώτη μας συνεδρίαση είναι το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό η ψηφοφορία επ' αυτών θα πρέπει να γίνει στις 12 Ιουλίου των τροπολογιών για τον προπολογισμό δηλαδή. Και δεν θα έχουμε την ε, πρόταση του Συμβουλίου, θα ψηφίσουμε μόνο το σχέδιο προπολογισμού της Επιτροπής. Και αν μετά χρειαστεί να γίνουν αλλαγές, ήδη ως εισηγήτρια μου δώσατε εξοδότηση να δράσω εκ μέρους σας και να κάνω περαιτέρω προσαρμογές αν χρειάζεται. Προθεσμία λοιπόν για τροπολογίες επίσης πολύ μικρή για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Ιούλιο. Πρέπει λοιπόν η προθεσμία να λήξει στις 6 το απόγευμα της 22ης Δευτέρας τρέχοντος. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τουλάχιστον η, κυρία Μπρέσο από τους Σκιώδης, οπότε θες να πεις κάτι, παρακαλώ. Καταρχάς ευχαριστώ. Ήθελα να σας συγχαρώ, διότι η πρόταση γνωμοδότησης ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει συμπεριλάβει και όλες τις προτάσεις για πιλωτικές δράσεις που είχαν προτείνει διάφορες πολιτικές ομάδες και νομίζω ότι γενικώ υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θέλουν να αυξήσουν τη σχέση με τους πολίτες, ε, να εκφράζονται περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες. Συμφωνούμε λοιπόν με τη γνωμοδότηση και τις τροπολογίες, τις σκεφτόμαστε. Αν κατάλαβα καλά, βέβαια δύο μέρες έχουμε στη διάθεσή μας για να δούμε το ενδεχόμενο ε, να προσθέσουμε και κάτι για ένα διαρθρωμένο διάλογο με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ε, με κινήματα που ασχολούνται εν γέννη με ευρωπαϊκά θέματα, όχι συγκεκριμένα που είναι λίγο παραμελημένη. Δηλαδή υπάρχει ο διαρθρωμένος διάλογος συνήθως, αλλά συνήθως γίνεται για κάποια συγκεκριμένα θέματα. Αλλά, για παράδειγμα, γενικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει διαρθρωμένος ε, διάλογος με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Καταρχάς, λοιπόν, το λέω σε εσά ε, ως πρόεδρο, Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε ίσως να θίξουμε, διότι υπάρχει μια ad hoc ε, εξουσιοδότηση στο συνάδελφο Βαρκάλσελ εκ μέρου του Προέδρου, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Ε, το προβλέπει ο κανονισμός, αλλά ποτέ δεν ε, έγινε κάποια απόπειρα επ' αυτού. Θα προτείνω λοιπόν ίσως κάποια μικρή φράση που θα υπενθυμίζει το θέμα αυτό ο διαρθρωμένος διάλογος να γίνεται και για μεγάλα θέματα και να μην γίνονται απλώς για κάποια συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένη νομοθεσία. Και ίσως εμείς να είμαστε αρμόδιοι να το θίξουμε ως Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων που έχει μια πιο ευρύτερη εικόνα των πραγμάτων. Αυτή είναι η μόνη παρατήρηση. Κατά τα λοιπά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω η παρατήρησή σας ήταν πάρα πολύ σημαντική και σοβαρή. Μπορούμε να το κλείσουμε λοιπόν το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να αναφέρω και το εξής. Δεν έκανα τις ανακοινώσεις της Προέδρου για τις αποφάσεις των συντονιστών σήμερα το πρωί και είναι και αρκετά σημαντικές διότι περιλαμβάνουν όλα τα σημαντικά έγγραφα τα οποία σκοπεύουμε να συντάξουμε ε, για την Επιτροπή ε, θέλει να πει κάτι, για τον προπολογισμό θέλει να πει κάτι που η Επιτροπή σήμερα σας ξεχνάω συνέχεια. Λοιπόν, συστάσεις των συντονιστών. Όσον αφορά τις εργασίες μας για το μέλλον της Ευρώπης, ε, συμφωνήσαμε να καταρτιστούν μια σειρά από έγγραφα εργασία για οκτώ θέματα και σήμερα ε, λήφθησαν αποφάσεις ε, για τους ε, βασικούς εισηγητές, δόθηκαν στις πολιτικές ομάδες. Επομένως τώρα περιμένουμε να μας πούν οι ομάδες όλες τις πληροφορίες για πιθανούς σκιώδεις εισηγητές σε όλες αυτές τις εκθέσεις και επίσης και συγκεκριμένα ονόματα ε, για αυτούς οι οποίοι θα αναλάβουν τα έγγραφα. Τώρα, για τις κοινωνικές ε, πτυχές ε, του παρόντος πλαισίου είναι η η αρμόδια μαζί με το EFTD για την παγκοσμιοποίηση το ΕΛΚ σε συνεργασία με τους φιλελευθέρους, για την Νομισματική Ένωση οι Σοσιαλδημοκράτες και το ΕΛΚ, για την άμυνα το ΕΛΚ οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και για τα οικονομικά της Ένωσης το ΕΛΚ και οι Σοσιαλιστές πάλι. Νόμιζα για την άμυνα ήταν άλλη, αλλά εσείς είστε ικανοποιημένοι. Έτσι αποφασίσετε. Έλκη και σοσιαλιστές για την άμυνα. Εντάξει, σοσιαλιστές και έλκη θα συνεργαστείτε. Για την ηθαγένεια, φίλε ελεύθεροι με τους πρασίνους και για ε, τη δομή και τη μέθοδο εργασία του Συμβουλίου, το ECR με τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και ε, για την ολοκλήρωση πράσινη. Επομένως, εδώ έχουμε ε, τις ομάδες. Ε, θα χρειαστούμε τα ονόματα και τους κοιόδης εισηγητές ε, όταν δεν έχετε εισηγητή. Συμφωνήσαμε επίση να διοργανωθεί μία ακρόαση για την αναθεώρηση του κανονισμού για το καταστατικό και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων. Αποφασίστηκε να γίνει η ακρόαση αυτή τον Ιούλιο στι 12 Ιουλίου και ο στόχο είναι να ε, χρησιμοποιηθεί για το προπαρασκευαστικό έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όπω μα επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια σκοπεύει να ε, καταθέσει νομοθετική πρόταση εντό του έτου αργότερα αργότερα βέβαια. Ε, έχουμε λοιπόν τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων και όσον αφορά την ημερήσια διάταξη θα το δούμε αύριο όταν θα έχουμε και τον τελικό κατάλογο για την ημερήσια διάταξη ε, του Ιουλίου, να δούμε πόσους μπορούμε να προσκαλέσουμε και εκπροσώπους πολιτικών ομάδων, αν μπορεί να γίνουν όλα μια φορά τον Ιούλιο ή αν θα πρέπει να χωριστεί συνεδρίαση στα δύο, να γίνουν δύο συνεδριάσεις ε, και να συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο, ε, για τις 4 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση θα γίνει ε, στις 12 Οκτωβρίου για το μέλλον της Ευρώπης και ένα τελευταίο θέμα, η ακρόαση που προβλέπεται για το δεύτερο εξάμεινο για τις ταγματικές ε, συνέπειες των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων της Λευκής Βέβλου για την Ένωση θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου. Επίσης συμφωνήσαμε ότι οι πολιτικές ομάδες θα στείλουν στη Γραμματεία προτάσεις για εμπειρογνώμονες ε, που θα προσκληθούν μέχρι την 5η 29 Ιουνίου. Συνολικά τρεις. Δεν μπορούμε να έχουμε παραπάνω. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση λοιπόν, ε, θεωρώ ότι οι συστάσεις των συντονιστών εγκρίνονται από την Επιτροπή. Επίσης, Συνήθως σας ενημερώνω για τα όσα συνέβησαν και που συμμετείχα για το Brexit. Είχαμε μία συνεδρίαση της Διευθύνουσας Επιτροπής ε, την 3η 13 Ιουνίου στο Στρασβούργο με παρουσία και του Μισελ Μπαρνιέ και μας παρουσίασε τις ε, εξελίξεις και την πρόοδο που έχουμε στην όλη διαδικασία ε, μας επανέλαβε με ποιο τρόπο θέλει να συνεργαστεί στο Ευρωπαϊκό, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διάφορες ε, διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, τους διάφορους κύκλους. Ε, ε εχθές ε, συναντήθηκε με τον David Davis, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια προσαρμογή στο κύκλο αυτό. Μπορεί να αλλάξει κάτι λοιπόν σε αυτό το κύκλο διαπραγματεύσεων. Ε, θα τα δούμε αυτά στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει σχετικά σύντομα. Αυτά λοιπόν από πλευράς μου. Επόμενη συνεδρίαση στις 12 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ πέρα τη συνεδρίαση.